Good morning to you all. I think that we... Καλημέρα σας. Νομίζω πριν να ξεκινήσουμε. Την εξέταση των υποψηφίων. Ιδίως να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπρένινγκ Μαγερό, ο οποίος έχει ήδη αναμείνει αρκετή ώρα. Έχουμε αργήσει. Ζητώ συγγνώμη και εγώ ίδια και βεβαίως εκ μέρους των μελών της Επιτροπής για αυτή την καθυστέρηση και καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας. Η σημερινή συνεδρίαση όπως ενημερωθήκαμε με εγκύκλιο που διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη περιλαμβάνει μία ώρα μια χρονοδιρίδα μια ώρας για κάθε υποψήφιο. Έχουμε έξι υποψηφίους που έχουν υποβάλει την αίτησή τους και ως γνωστόν η Προεδρία έχει ασχοληθεί με την πρώτη διοικητική φάση της ε, εξέτασης αποδεκτού των ψηφιότητων, παραδεκτού μάλλον, ενώ εμείς έχουμε την ε, αρμοδιότητα να επιτρέψουμε στους έξι έγκυρους υποψηφίους να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. Μετά θα καταλήξουμε σε ψηφοφορία στην Ολομέλεια, η οποία θα διασφαλίσει την ε, συγκατάθεση ή όχι σε σχέση με τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν. Και αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίω από την ψήφο των Ευρωβουλευτών. Θα προχωρήσουμε ακούγοντας με αλφαβητική σειρά τους υποψηφίους και θα δώσουμε στον καθένα την ευκαιρία να κάνουν μια αρχική ομιλία έπειτα ούτως ή άλλως έχουμε δώσει την ευκαιρία να εκφραστούν οι υποψήφοι έχοντας αποστείλει γραπτές ερωτήσεις, γραπτές ερωτήσεις τις οποίες απήντησαν και έχουν ήδη δημοσιευθεί και μετά από αυτές τις παρουσιάσεις θα ακολουθήσουν ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών με έναν πρώτο γύρο ώστε να ακούσουμε πρώτα τους συντονιστές και να ακολουθήσουμε και κάποια ιεραρχία εδώ πάντοτε ανάλογα με την ε, σύνθεση και την ισχύ των ε, πολιτικών ομάδων. Και μετά θα προχωρήσουμε με τη μέθοδο Catch the Eye. Καλό λοιπόν τους συναδέλφους να σεβαστούν τα χρονικά περιθώρια, διότι στο πλαίσιο της σημερινής ημέρας πρέπει να ακούσουμε και τους έξι υποψηφίους. Πάνω απ' όλα πρέπει να δείξουμε σεβασμό προς τους υποψηφίους αυτούς αλλά και να φροντίσουμε να περάσει το μήνυμα το οποίο να λαμβάνουμε την ευθύνη. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον πρώτο μα υποψήφιο. Και πάλι του ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Όμως, όπως και σε όλου τους άλλους υποψηφίου θα του δώσουμε το χρόνο που του έχουμε ήδη ε, ορίσει. Παρακαλώ. Thank you, Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας προσφέρω την υποψηφιότητά μου. Βεβαίω θα μπορούσα να σας κάνω την παρουσίασή μου στα Ολλανδικά, αλλά νομίζω ότι ως δημοσιολαβητής είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορώ με πιο άμεσο τρόπο να επικοινωνήσω. Οπότε και για αυτό θα σας αναπτύξω τα επιχειρηματά μου ή στα Αγγλικά. Είναι μεγάλη μου τιμή να σα παρουσιάσω την υποψηφιότητά μου για την θέση του Ευρωπαίου Δημοσιολαβητή και έτσι που θα απαντήσω στι τρεις αυτέ ερωτήσει, Η πρώτη πρώτη είναι ποιο είμαι. Η δεύτερη τι αντιπροσωπεύω και τρίτον γιατί κατεβαίνω ως υποψήφιος. Πρώτον, ποιο είμαι. Την τελευταία τριακονταετία έχω αποκτήσει εμπειρία ως δικαστής και αντιπρόεδρος του εφετείου και νομικός αποφύτησα από το Λάιντεν και ειδικεύομαι στην ε, επιδιαιτησία, διαμεσολάβηση και επίλυση επιδίκων διαφορών. Επί 8 χρόνια είχα θέσει το δημοσιολαβητή στη χώρα μου και όταν ξανακατέβηκα για υποψήφιος συνεκέντρωσα την ε, συμφωνία όλου του σώματος εκτός από το κόμμα του Βίλντες. Θα πρέπει να σέβεται πιστεύω και το κοινό και τον κόσμο και του θεσμού οπότε τελευταία μου είπαν ότι όχι μόνο είμαι ο μαχητής για τον κόσμο, αλλά επίσης ότι έχω εμβρεθεί γνώση των υποθέσεων και ότι είμαι πάρα πολύ φιλότιμος, δουλευταράς και ότι έχω ηθική ακυριότητα. Η απλή γλώσσα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το έργο μου. Μέσω των ΜΜΕ έχω συνεχή επαφή με τους πολίτες, με συνεντεύξεις και γράφω μια φορά τη βδομάδα στην ε, πιο δημοφιλή εφημερίδα μας και σε μέσα από μέρες πρόκειται να σας διαβάσω με λιγότερο ταχυδρομείο κάποια από τα άρθρα μου. Θεωρείτε ότι διαμορφώνω την άποψη στη χώρα μου όσον αφορά την χρηστική κυβέρνηση και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και έχουν πάρα πολλές ε, περιπτώσεις που μου εμπιστεύονται και υποθέσεις οι πολίτες γιατί με, ακριβώς γιατί με εμπιστεύονται. Όσον αφορά τους καταγγέλλοντες και αυτοί με εμπιστεύονται όπως επίσης και τα ΜΜΕ και ήμουν ο βασικός ομιλητής όταν εκλέξαμε τον δημοσιογράφο της χρονιάς για το 2012. Τη ίδια χρονιά επίσης είχαμε την ετήσια συνάντηση των δημοσιογράφων που κάνουν ρεπορτάζ κοινοβουλίου στη Χάγη. Επίσης, ο φορέας των δημοσιογράφων που κάνουν τις έρευνες, επίσης με έχουν καλέσει να δημοσιολαβήσουν όταν θέλανε να αναβαθμίσουν την ε, διαφάνεια στο δημόσιο. είμαι καινοτόμος, είμαι δημιουργικός, είμαι αποφασιστικός, χωρίς να είμαι όμως βάναυσος. Οπότε η, η θέση του διαμεσολαβητή για μας είναι κάτι στο οποίο έχουν όλοι προσβασιμότητα και οι πολίτες και οι δημόσιες υπηρεσίες. Το Υπουργείο Εσωτερικών οργάνωσε μια μεγάλη κλίμακα ε, ε, έργο, ούτως ώστε να βελτιώσει τα πράγματα και έτσι προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τις ε, διαδικασίες ε, τις νομικές και 60% των υποθέσεων τελικά δεν καταλήγει σε ε, προσφυγή στο δικαστήριο, ή σε μήνυση. Αυτό ήταν επομένω το όραμα που ήθελα να ολοκληρώσω και έτσι η θέση του διαμεσολαβητή στη χώρα μας ήλκησε την προσοχή και έχουμε επομένως συνεργασία με χώρες όπως Τσεχία, Ρουμανία, Βουλγαρία Εσπανία και Σερβία. Επίσης, σε Σουηδία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο, δύο μεσολαβητές, ε, ενδιαφέρθηκαν να μάθουν τη δική μας μέθοδο. Και πρόσφατα ήρθε στο γραφείο μας ο Σουηδός με το προσωπικό του για να μάθει τη μέθοδό μας. Και πρόσφατα κάλεσα και συμβούλευσα εκπροσώπους της ε, Κοπενχάγης για το πώς θα βελτιώσουν εκεί τα πράγματα και έτσι και έτσι πώς θα μεταλαμβαρέσουμε τέλος πάντων αυτό που κάνουμε. Οι δε συναδελφοί μου με εξέλεξαν ως ε, πρόεδρο του Φορέα των Ευρωπαϊκών Συμμελοβητών. Δεύτερη ερώτηση τώρα. Γιατί διάλεξα να κάτω υποψήφιο και τι εκπροσωπώ. Θεωρώ ότι ο Δημοσιολαβητή αποτελεί την ανθρώπινη διάσταση ακόμα και στα πιο τεχνοκρατικά και περίπλοκα ζητήματα. Στη δημόσια διοίκηση, η ανθρώπινη διάσταση πρέπει να φορά δεν την προσέχουμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση. Δεν θα πρέπει να δίνουμε το βάρος στην νομική διάσταση. Ταυτόχρονα πάντως θα πρέπει να γνωρίζει νομικά ο υποψήφιος γιατί πρόκειται για περιπτώσεις όπως τη Σόλαφ, για τον Ντάλι, διαφάνεια, ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μου είναι βασικό για να δικαιωθούν αυτές οι υποθέσεις να πρέπει να γνωρίζει νομικά ο διαμεσολαβητής. Επίσης, για να είναι μετά, <coughs> Ε, δεν θα πρέπει να ακολουθεί τις απόψεις των συνεργατών του, θα πρέπει να πιστεύετε τη δική του άποψη. Οπότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια κωδικά για την διοίκηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένω όλα τα θεσμικά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης πολλές φορές χάνονται μέσα στην ζούγκλα της ε, πολυνομίας. Ο κύριος Διαμαντούρος αυτό το θέμα το θεωρώ ο της προτεραιότητας και ορθώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια όθηση σε ακριβώς αυτό το όραμα του κ. Διαμαντούρου. Επόμενο, το να αναζητήσουμε την ανθρώπινη διάσταση στις περίπλοκες υποθέσεις είναι δική μου φιλοδοξία. Θα πρέπει ο κόσμος να μην έχει αντιμετωπίσει ε, περίπλοκες διαδικασίες. Θα πρέπει να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματά τους. Για παράδειγμα, εάν κάποιος δεν λαμβάνει απάντηση εγκαίρως, θα πρέπει αυτό να διεκπεριώνεται. Θα πρέπει να δίνονται αιτιολογήσεις για τις αποφάσεις, πρακτικές αποφάσεις μεταξύ διαμεσολαβητή και αρχών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στο να ξεβρίσκονται λύσεις αυθημερών ή την ίδια εβδομάδα ή τον ίδιο μήνα, εάν χρειάζεται. Θα πρέπει επομένω να μην είναι γραφειοκράτης ο διαμεσολαβητής και ούτε είναι αυτό αυτός σκοπός διεκπαιρέωση των καταγγελιών και παράπονα. Από την άλλη μεριά όμω. αυτά, αυτά τα παράπονα καταγγελίε μπορούν να μα ενημερώσουν για το τι είδου διαρθωτικά δομικά προβλήματα ε, είναι η ρίζα του κακού. Οπότε και έτσι θα πρέπει με συστημικού χαρακτήρα έρευνε να βλέπουμε πώ μπορούμε να επιφέρουμε βελτιώσει. Οπότε και τα θεσμικά όργανα μπορούν να διδαχθούν από αυτέ τι καταγγελίε Και με αυτή τη μέθοδο θεωρώ ότι πέτυχα να επιφέρω βελτιώσεις. Όπως η συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων, ε, πάροχη αποζημιώσεων, ε, διατύπωση αποφάσεων σε κατανοητή απλή γλώσσα και επίσης περισσότερη σύνδεση του δημοσιοδητή με τα ΜΜΕ. Έτσι, μπορεί να συμφιχθούν περισσότερε σχέσει με τους πολίτε και ιδίω με του νέου. Πολύ σημαντικό θέμα επίση είναι ποιες καταγγελίες δεν φτάνουν διαμεσολαβητή από τους πολίτες. Θα πρέπει ομένως ο διαμεσολαβητής εκείνος να αναζητεί τις καταγγελίες. Τώρα, για ποιο λόγο ακριβώς κατεβαίνει υποψήφιος. Η γυναίκα μου γεννήθηκε στην Τσεχοσλοβακία και μετά την άνοιξη της Πράγας το 1968 ήρθε στις κάτω χώρες. Και εν μέρη, λόγω της ιστορίας της ζωής της γυναίκας μου, για μένα η Ευρώπη δεν είναι ένα νεκρογράμμα. Η ε, ειρήνη και ελευθερία είναι η, καρδιά της Ευρώπης, οπότε αυτό είναι το μέλλον το κοινό μας. Δεν πρόκειται για απλά έναν θεσμό. Αυτό το οποίο θέλω είναι να υπάρχει περισσότερη δικαιοσύνη στην αντιμετώπιση των πολιτών από πλευρά θεσμικών οργάνων. Οι έρευνε που έχω διεξαγάγει Βλέπετε αυτό το έντυπο και υπάρχει στο ίντερνετ. Ε, έκανε κάτι στο συμπεραστό ότι τα νομικά συστήματα είναι περιπλοκά και πολλές φορές οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν γιατί η ζωή τους επηρεάζεται από τις ενέργειες της διοίκησης. Αυτό θα πρέπει να μην το ξεχνάμε και ότι η εμπιστοσύνη είναι το πιο κρίσιμο, το πιο σημαντικό. Και υπάρχει εμπιστοσύνη όταν έχουμε δικαιοσύνη και όταν έχουμε διαφάνεια και για την διαφάνεια. Όντως υπάρχουν κάποια συμφέροντα που επιβάλλουν περιορισμού στη διαφάνεια. Όμως κατά τη γνώμη μου η διακυβέρνηση Ευρωπαϊκή θα πρέπει να είναι ανοιχτή διακυβέρνηση. Απλώ τα πράγματα υπάρχουν κάποια, κάποια όρια του απορρίτου γιατί ο κόσμο θέλει να καταλαβαίνει τι γίνεται. Οπότε και η Ευρώπη θα πρέπει να παράσχει ενημέρωση και να υπάρχει έτσι κατανόηση. Έχουμε το κανονισμό 1049 που θα πρέπει να είναι πάνω-πάνω στην ε, ημέρηση διάταξη. Κάθε νομοθέτη επίσης θα πρέπει να δίνει τη μάχη του συνέχεια ο διαμεσολαβητής για την χρηστή διακυβέρνηση και για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Θα πρέπει να φροντίζει επίσης τα θεσμικά όργανα να ε, χειρίζονται τις υποθέσεις των πολιτών δίκαια. Ε, βέβαια δεν είναι όλε οι αποφάσει θετικέ, πολλές φορές είναι απογοητευτικέ οι αποφάσει τη διοίκηση για του πολίτε, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την ε, δίκαιη διεκπαιρέωση, ακόμα και στι αρνητικές ε, αποφάσει. Διαφάνεια και δικαιοσύνη. Αυτό είναι κάτι που με αγγίζει και με συγκινεί βαθιά και ω άνθρωπο και ω πανεπιστημιακό και ω διαμεσολαβητή. <coughs> Οπότε και αυτό είναι το βασικό μου κίνητρο και ε, για να γίνω νέο Ευρωπαίο Δημοσιολογητή. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Ευχαριστούμε κύριε Μπρένιγκ Μάιερ. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας και για το ότι σεβαστήκατε και το χρόνο. Ελπίζω τώρα και οι βουλευτές να κάνουν το ίδιο. Ο κύριος Γιάρη έχει πρώτο λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Μπρένιγκ Καλή αρχή όπως είπε και η Πρόεδρο, στηρίσατε το χρόνο ομιλίας. Και ελπίζω ανάλογα να κινηθείτε και αν γίνετε διαμεσολαβητής. Έχω κάποιες ερωτήσεις για εσάς. Τη σημαντικότερη είναι η πρώτη γιατί συζητιέται πάρα πολύ και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι το θέμα της ανεξαρτησίας. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς θα ορίζατε την ανεξαρτησία ποια είναι τα όρια της ανεξαρτησίας, αν σας υποστηρίζει κάποιος και επιπλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ε, διαφορετικές ε, καταστάσεις. Η Γερμανία δεν έχει διαμεσολαβητή. Άλλες χώρες έχουν ε, πολύ έντονο τέτοιο χαρακτήρα στο θεσμικό αυτό όργανο και επίσης ακούω πως θα έπρεπε να είναι ένα ουδέτερο μέλος του Κοινοβουλίου αυτό θα ήθελα να πούμε η Σουηδία και η Ολλανδία. Θεωρείται σωστό να είναι ταυτόχρονα βουλευτής ε, ο διαμεσολαβητής. Κατόπιν, άλλο ερώτημα. Ποια είναι για σας τα τρία σημαντικότερα πράγματα. Με τι θα ασχοληθείτε αν γίνετε διαμεσολαβητής κατόπιν για την δημοσιότητα του αξιώματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θεωρώ πως ε, θα πρέπει να έρθει πιο κοντά στους πολίτες ο θεσμός αυτός. Οπότε το ερώτημα είναι πώς φαντάζεστε ε, ότι θα μπορέσει να έρθει πιο πολύ στη δημοσιότητα ο Διαμεσολαβητής. Επόμενο θέμα, χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πώς βλέπετε το ζήτημα ότι δεν ε, είναι τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικαίου η χάρτα, αλλά ένα επιπλέον ε, πρωτόκολλο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις, ε, πάρα πολλές αναφορές για, που αγγίζουν το ζήτημα αυτό. και είναι βέβαια και το ζήτημα τη αρμοδιότητα τη ε, δική μας, που δεν επαρκεί. Και τελευταίο ερώτημα. Ποια είναι η σχέση, θεωρείτε, της υπηρεσίας σας και της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πώς το βλέπετε να διαμορφώνετε συγκεκριμένα αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, κύριε Γιάρ. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Μπέρμαν, του Σοσιαλιστέ. γιατί δεν είναι εδώ ο συντονιστής. Εντάξει, έχετε το λόγο. Ένα ερώτημα θα ήθελα να θέσω. Ποια θεωρεί ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ εθνικού και ευρωπαίου διαμεσολαβητή και πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη διαφορά στους ρόλους, πώς θα εκπληρώσει το ρόλο του. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια διαφορά. Ευχαριστώ. Άουκεν. Ευχαριστώ κύριε Μπρεν και ευχαριστούμε για την ε, επίσκεψή σας εδώ. Να προσθέσω στην ερώτηση του κύριου Μπέρμαν το εξή. Μιλούμε για την προβολή και ελπίζω να καταλαβαίνετε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά με το τι γίνεται εδώ και το Εθνικό Κοινοβούλιο και τους διαμεσολαβητές του. Εγώ ήμουν 20 χρόνια βουλευτής στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Ξέρω πόσο δύσκολη είναι αυτή η προσπάθεια. Ξέρετε λοιπόν πώς μπορεί να γίνει αυτό χωρίς απλώς να παραμένουν όλα αυτά ευσεβείς πόθη. Και ως προς την ερώτηση του κυρίου Μπέρμαν. Οι θεσμοί και τα θεσμικά όργανα που δέχονται επικριτικά σχόλια το ίδιο το κοινοβούλιο. Ε, πώς μπορεί αυτό να συγκρίνεται με τις κάτω δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχετε ε, λοιπόν εμπειρία από πραγματικά έτσι, σκληρά θεσμικά παιχνίδια και τι πρέπει να κάνει κανείς για να κερδίσει πολιτική στήριξη. Όχι προσχώρηση ή κομματική στήριξη, αλλά πολιτική ισχύ, πυγμή. Και ως προς την ανεξαρτησία, σας θεωρώ ανεξάρτητο υποψήφιο δημοσιολαβητή και βάσει του νόμου για την καλή διοικητική συμπεριφορά και για την ανεξαρτησία. Δεν είναι απλώς μια αίσθηση, είναι σαφές αυτό. Υπάρχει νόμος για το τι είναι καλή χρηστή διοίκηση και αναφέρεται εκεί ορισμό της ανεξαρτησίας. Για τη διαφάνεια όμως. Η διαφάνεια είναι ένας διαρκής αγώνας που δίνουμε σε αυτό το σώμα. Και ακόμη και για την περίπτωση των εκλογών η διαφάνεια χρειάζεται ακόμα περισσότερο από τις άλλες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι απλό. Δεν είναι απλό να υπάρχει διαφάνεια όταν ε, βλέπουμε εδώ να μην την προωθεί η ίδια η Προεδρία του Κοινοβουλίου. Τώρα όμως είστε στην Επιτροπή Αναφορών. Αναφέρατε κι εσείς ο ίδιος το 249. Θα υπάρξει κάποιο κανονισμός για την καλή διοικητική συμπεριφορά όχι ένας ε, δεσμευτικός και άκαμπτος κανονισμός, αλλά νομίζω ότι πραγματικά χρειάζεται κανονισμός εδώ. Προς τα θεσμικά όργανα για την καλή δίκηση, τη χρηστή δίκηση. Και να το συνδυάσω αυτό και με την ε, διαφάνεια. Η σύμβαση του όρχους δεν βλέπω να γίνεται σεβαστή. Έχω πολύ λέγα τέτοια δείγματα μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Δεν βλέπω να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια. Τι ιδέες έχετε εσείς για το πώς θα μπορούσαμε να το υλοποιήσουμε αυτό, να περάσει στο, γενό, στο γονότυπο των, ε, των, των διοικητικών υπαλλήλων του βηματός μας. Περισσότερη διαφάνεια, περισσότερο ανοιχτό πνεύμα. Αυτό χρειάζεται. Και αναφέρατε πάρα πολύ το πόσο σημαντικό είναι να έχει κανείς γνώσει νομική. Είστε δικηγόρος, είσαστε πολύ καλό υποψήφιο. even if he's not a lawyer. παρά το ότι δεν είναι νομικός ο κ. Διαμαντούρος, είναι πολύ υψηλού επίπεδου διαμεσολαβητής. Σας ευχαριστώ, κ. Σαλαβράκος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, θεωρώ ότι και σοβαρό βιογραφικό είχε ο υποψηφιός μας και σοβαρότητα στην ανάπτυξη των ε, θέσεών του. Ε, εγώ δεν θα πω πολλά. Ξέρετε ότι είμαι από εκείνους που στηρίζω το θεσμό του Ομπούσμαν και ο προβληματισμός μου είναι κατά πόσον θα μπορέσουμε στο θεσμό αυτό να δώσουμε μία εκτελεστότητα στις αποφάσεις του Ομπούσμαν. Διότι μέχρι τώρα, όπως γνωρίζετε, οι αποφάσεις του Ομπούσμαν δεν είναι εκτελεστές, ε, βασίζονται στο σεβασμό προς τον θεσμό τον οποίο επιδεικνύουν τα κράτη, αλλά αυτό δεν αποτελεί νομική δέσμευση. Προς την κατεύθυνση αυτή θα ήθελα να ακούσω τις σκέψεις και τις προτάσεις τις οποίες θα ε, έκανε ο υποψήφιος σε περίπτωση που καταλαμβάνει τη θέση. Ευχαριστώ πολύ. Thank Ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσεστερ. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Μπρένικ Μάιερ. Ε, Χάρηκα που σας γνώρισα. Ελπίζω να έχετε δυνατή μνήμη και να σημειώνετε κιόλας, γιατί έχω κι εγώ πολλές ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι κάπως γενική. Και θα ήθελα να δω έτσι την οπτική σας γωνία ως ανεξάρτητος αξιωματούχος. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να αποκατασταθεί εν μέρη ε, η εικόνα των πολιτικών και αν είναι δουλειά αυτή του διαμεσολαβητή. Δεύτερον, με τη δική σας την εμπειρία, ε, θεωρείτε πως πολιτικοί ή αξιωματούχοι ε, συνεργάζονται περισσότερο, συνεργάζονται αρκετά περισσότερο ή λιγότερο με τον διαμεσολαβητή. Γιατί ξέρετε, οι αξιωματούχοι ε, και οι υπάλληλοι δεν ε, εκλέγονται και δεν ε, έχουν πίεση. Και μετά σκέφτομαι και το βασανιστήριο που περνάτε αυτή τη στιγμή. Πείτε μας ποια ήταν η διαδικασία που περάσατε για να γίνετε διαμεσολαβητής ε, στην Ολλανδία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τσίτσιστερ. Ε, πρέπει νομίζω να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μπρένινγκ Μάιερ να απαντήσει τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και μετά ξεκινάμε το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύ καλές ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να τις απαντήσω όλες. Αλλά μετά θα μπορέσω να σεβαστώ το φραγκόριο. Και αυτό πρέπει να κάνει κάθε φορά ο διαμεσολαβητής, πρέπει να σέβεται τα, τις προθεσμίες. Ναι, με ρωτήσατε τώρα κύριε Γιάρ για την ανεξαρτησία του του. Θεωρώ πως είναι πάρα πολύ σημαντική ανεξαρτησία και η απάντηση αυτή νομίζω μπορεί να συνδυαστεί με την απάντηση στην ερώτηση του κυρίου Τσίτσεστερ ο οποίος ε, ρώτησε ποια ήταν η διαδικασία στην Ολλανδία. Στην Ολλανδία, στις κάτω χώρες. Ε, υποβάλλει κάποιος αίτηση και υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και προτείνουν αυτοί τρία άτομα στο Κοινοβούλιο και θεωρώ πως επιλέγουν υποψηφίους με βάση τις ικανότητές τους και μετά είναι ζήτημα του εάν θέλει κανείς άντρα, γυναίκα τα λοιπά Και ίσως και άλλα ζητήματα. Και δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτή τη διαδικασία. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που ετέθη ήταν το ζήτημα της δημοσιότητας ε, του διαμεσολαβητή. Το πώς θα γίνει πιο γνωστό, το θεσμικό όργανο ε, σε, στα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους. Κοιτάξτε, το ίδιο ισχύει και στην Ολλανδία. Ήταν άγνωστος ο διαμεσολαβητής. Χρειάστηκε λίγο χρόνος, αλλά σήμερα ξέρουν όλοι ποιος είναι ο διαμεσολαβητής και τι κάνει, οπότε εγώ θεωρώ πως έχω την εμπειρία και βεβαίω, κυρία Άουκεν, στην Ευρώπη είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εάν επικοινωνεί κανεί σε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ολλανδικά, μπορεί νομίζω να πείσει το, τον κόσμο και να μιλάει τη γλώσσα του απλού ανθρώπου αν μπει στο ίντερνετ, ανεβάσει κάποιες ταινιούλες. Μπορεί ε, να επιτελέσει αυτό το ρόλο. Και βέβαια πρέπει και κάποια τεχνικά ζητήματα να μεταφραστούν σε καθημερινή γλώσσα και να εξηγήσουμε το γιατί είναι σημαντικό παραδείγματο χάρη να έχουμε διαφάνεια, γιατί να έχουμε ανθρώπινα δικαιώματα κτλ. Νομίζω πως ένα από τα πλεονεκτήματα του διαμεσολαβητού είναι πως δεν σχετίζεται άμεσα με τον νόμο. Η δουλειά του είναι η δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και σε αντίθεση με ένα δικαστήριο μπορεί να εφαρμόσει σε κάποιες περιπτώσεις να αναπτύξει κάποια επιχειρήματα για να πείσει το γιατί καταλήγει σε μια αρνητική απόφαση για αυτό κάτι το οποίο έκανε η Και στην περίπτωση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντικό να πείθουμε τον κόσμο. Και ξεκίνησα να λέω πως είμαι ειδικό στις διαπραγματεύσεις, ε, στη διαμεσολάβηση και στην επίλυση κρίσεων. Γιατί, αν με ρωτήσετε, αν χρειάζεται περισσότερες αρμοδιότητες, ο διαμεσολαβητής, εάν πρέπει να έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις. Όχι θα έλεγα πως ε, τα ισχυρότερα του όπλα είναι τα επιχειρήματά του, οι κανόνες, τα ανθρώπινα αλλά το πώς, το πώς επιχειρηματολογεί δεν πρέπει να είναι χαρτούρα. Πρέπει να έρχεται σε επαφή με την διοίκηση. Εγώ είχα πολλές επαφές με τη διοίκηση και τώρα έρχονται στο γραφείο μου και μου λένε έχουμε ένα πρόβλημα. Ε, γιατί ο χύψη πολίτης ε, έχει κάποιο ζήτημα. Και με την εμπιστοσύνη των ε, πολιτών. Και αυτό ήταν και το αντικείμενο της έκθεσής μου το 2011. Και πολιτικοί και ε, μέλη της διοίκησης ήταν πάρα πολύ ικανοποιημένοι με την άποψή μου. Και εάν ρωτήσετε κύριε Γιάρ για τα τρία σημαντικότερα ζητήματα για εμένα θα έλεγα, δημοσιότητα. Το να εξηγούμε, το να πείθουμε τον κόσμο το γιατί χρειάζεται ο διαμεσολαβητής. Δεύτερον, πρέπει να δράμε τρόπο γρήγορο και άμεσο, δεν και λύς διαδικασίες, οπότε δεν θα πρέπει να είναι γραφειοκρατία, εάν θέλετε, και πρέπει βέβαια να έχουν πολύ καλές επαφές με τη δημόσια διοίκηση και ο κύριος Τσίτσεστερ ρώτησε ε, το εάν κάποιοι συνεργάζονται περισσότερο και λιγότερο. Ναι, κάποιοι συνεργάζονται λιγότερο πράγματι, αλλά ε, θα πρέπει να ξεκινήσω με αυτούς που συνεργάζονται περισσότερο, θα έλεγα, με τις διοικήσεις και τους πολιτικούς εκείνους που είναι πιο συνεργάσιμοι. Γιατί αυτοί μπορεί να επιφέρουν την αλλαγή να δείξουν το τι γίνεται αν ε, επιδεικνύει κανείς διαφάνεια και δικαιοσύνη. Και έτσι εδώ στην Ολλανδία έχω μια ομάδα ε, υπαλλήλων και πολιτικών ε, που με υποστηρίζουν και λένε δείξε μας το δρόμο και μετά θέλουν και άλλοι να ακολουθήσουν σε αυτή την πορεία. Και άρα έρχομαι στο ερώτημα αν υπάρχει ουσιαστική διαφορά μεταξύ Ευρωπαίου και εθνικού διαμεσολαβητή. Ναι, μία βασική διαφορά είναι πως ο Ευρωπαίος διαμεσολαβητής εργάζεται σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο. Το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ευρωπαϊκά θεσμικά οργάνωση είναι σε ένα πιο αφηρημένο επίπεδο και αυτό σημαίνει πως ε, οι περισσότερες περιπτώσεις είναι περιπτώσεις τελικά για τον εθνικό διαμεσολαβητή. Οπότε οι επαφές με τον εθνικό διαμεσολαβητή είναι πάρα πολύ σημαντικές και άρα οι πολίτες ε, μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Αλλά από την άλλη θεωρώ πως στην Ευρώπη μπορούμε να βρούμε κάποια πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με τη διαφάνεια, με τη δικαιοσύνη που μπορεί να χρησιμοποιήσει νομίζω θα έλεγα ο διαμεσολαβητής για να έρθει στο κοινό το μήνυμα του διαμεσολαβητή και να έχει την αίσθηση πως το κοινό προστατεύεται π.χ. ότι οι καταγγέλλοντες ε, έχουν την δυνατότητα να προσφύγουν ε, στον διαμεσολαβητή και θα τύχουν δικής μεταχείρισης. Νομίζω πως απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Ορίστε. Ναι, ναι, η σύμβαση του άρχους, ναι. Είναι τεχνικό το ζήτημα τώρα και για τον ε, διαμεσολαβητή το θέμα είναι αν πρέπει να μπει στην ερμηνεία της σύμβασης του άρχους ή αν μπορεί να πείσει πως οι βασικές ιδέες για τη διαφάνεια, για τη συμμετοχή μπορούν να εφαρμοστούν. Και στον τομέα αυτών θεωρώ πως από τη μία μπορώ να συνηγορήσω υπέρ της αγωγής ε, στοιχείων της σύμβασης του άρχου στη δουλειά του Δημοσιολαβητή, αλλά από την άλλη πως δεν υπάρχει κάποιο όριο στον διαμεσολαβητή για τα επιχειρήματα που θα χρησιμοποιήσει και λέτε πως ε, ακόμα και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου είναι κατά της διαφάνειας. Ε, εγώ θεωρώ πως δεν είναι πάντα αναγκαίο να μπλέξει κανείς ε, καυγά και διαφωνία. Βεβαίως αντιλαμβάνομαι πως η πολιτική καμιά φορά έτσι είναι. Αλλά από την άλλη ως διαμεσολαβητής, ως διαπραγματευτής έχω την ε, εμπειρία πως ε, μπορεί να επιτύχει κανείς στους στόχους του με καλό τρόπο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε να περάσουμε στο δεύτερο γύρο, κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Μπρίνκμαγερ. Μπρίνκμαγερ μάλλον. Δεν ήμουν εδώ για την αρχική σας ομιλία δυστυχώς, αλλά μιλήσατε για την ε, προβολή και τη διαφάνεια. Ξέρετε ότι το Κοινοβούλιο αναθεωρεί τον κανονισμό περί δημόσιας πρόσβασης στα έγγραφα. Σε ό,τι αφορά τα θεσμικά λοιπόν στοιχεία των αρμοδιοτήτων σα, τι ισορροπία πιστεύετε ότι μπορεί να βρεθεί μεταξύ πραγματικής και ουσιαστική λήψη αποφάσεων στα θεσμικά όργανα, αλλά και τη ε, ε, δυνατότητα τη κοινή γνώμη να ενημερώνεται. Για να υπάρχει σωστή ισορροπία. Οι άνθρωποι αισθάνονται απομακρυσμένοι από την Ευρώπη και τελείω ε, εκτό του παιχνιδιού. Πρόεδρο. Ο κύριο Γιάρκε πάλι, ω εκπρόσωπο του κυρίου Βαλέσα αυτή τη φορά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Βαλέσα δυστυχώς είναι σε μία ψηφοφορία. Μου ζήτησε να μεταφέρω μία ερώτηση. Mm. Στην ε, Ολλανδία υπάρχει διακριτική μεταχείριση πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εις βάρος ε, Πολωνών όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και αν σημαίνει κάτι τέτοιο ε, εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι. Σας ευχαριστώ αυτή ήταν τελευταία ερώτηση. Σας δίνω και πάλι το λόγο για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Κάσμαν για την κέρια ερώτησή σας για την πρόσβαση του κοινού, δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα και το κατά πόσο αυτή μπορεί να είναι ισόρροπη και συναρμοσμένη με την ανάγκη των ε, πολιτικών εθνών να έχουν και κάποια εμπιστευτικότητα στην χάραξη της πολιτικής, στη φάση χάραξης μάλλον της πολιτικής και την προετοιμασία των αποφάσεων. Νομίζω το θέμα αυτό είναι επίκαιρο και στην Ευρώπη και στις κατοχώρες. Χθε στις κατοχώρες έγινε συζήτηση για την πρόσβαση στα έγγραφα, τη διαφάνεια ε, και τη διαδικασία την πολιτική γενικότερα στη Χάγη άκουσα τους πολιτικούς και τα ανώτατα στελέχη να έχουν τη διάθεση σε ένα βαθμό τα έγγραφα να μένουν εμπιστευτικά. Ποιος είναι εδώ ο ρόλος του διαμεσολαβητή. Από τη μια ο διαμεσολαβητής μπορεί να έχει καθοριστικό ρόλο διότι να, μπορεί να γίνει ο κριτής της υπόθεσης αυτής βάσει των κανόνων διαφάνειας μπορεί να δει κατά πόσον τα κωδικοποιημένα έγγραφα θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται ή όχι. Μπορεί να παίξει λοιπόν το ρόλο του κριτή. Το θέμα είναι αν είναι αποτελεσματικό το ρόλο αυτό ή αν μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο που να του επιτρέπει να μεταφράζει τη φωνή του δικαίου, να είναι ο συνήγορος της εμπιστοσύνης του κοινού. Εγώ νομίζω ότι ο μεσολαβητή δεν θα πρέπει να επιλέγει ή το ένα ή το άλλο. Θα πρέπει να παίζει και του δύο ρόλου. Πολλέ φορέ ο διαμεσολαβητή πρέπει να είναι πολύ ακριβή σε αυτό το σώμα ή σε άλλα μέρη, λέγοντας ότι το τάδε το τάδε έγγραφο θα πρέπει να είναι προσβάσιμο για το κοινό και μάλιστα με σχετική ταχύτητα. Βλέπουμε οι δημοσιογράφοι να κινούν συνέχεια νομικές υποθέσεις για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα. Και αυτό ε, και χρονοβόρο είναι και κοστίζει και τελικά όταν κάποια στιγμή δημοσιοποιείται το έγγραφο δεν είναι καθόλου επίκαιρο. Η ανάγκη λοιπόν για, την, ε, για το άνοιγμα στο κοινό είναι κάτι που χρειάζεται σήμερα συνήθως, όχι αύριο ούτε μεθαύριο. Ε, πρέπει να είναι κανείς λοιπόν ταχύς. Και στη χώρα μου έχω προσκληθεί από τα αρμόδια υπουργεία στη Χάγη και για την Ένωση των Ανακριτών Δημοσιογράφων, ώστε να λειτουργώ ως διαμεσολαβητής μεταξύ τους, ως διαιτητής, όχι για νομικά ζητήματα, γιατί το νόμο το γνωρίζουν, γνωρίζουν τις διαδικασίες και τη δικονομία. Θέλουν να διαπραγματευτούμε για να δουν πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε σε καθημερινό επίπεδο την ανάγκη ενημέρωσης του κοινού, την ανάγκη ενημέρωσης των δημοσιογράφων και από την άλλη την ανάγκη προστασίας κάποιων συγκεκριμένων πληροφοριών και ουσιαστικά συμφερόντων. Συμφερόντων μιας δημοκρατικής πλευράς. Τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εάν κοιτάξουμε τη δικασία για την νομική συμβουλή για την νομική εμπειρογνωμοσύνη. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανεί στου πολίτε αυτό το επίπεδο τι γίνεται ακριβώ. Κατά την άποψή μου υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ των νομικών συμβουλών που θα πρέπει να δημοσιοποιούνται. Όμω, ε, ε καθώ είναι μέρο τη συζήτηση, έχουν και οι πολίτε την ανάγκη να συμμετέχουν σε αυτέ τι συζητήσει. Δεν είναι λοιπόν μόνο η διαφάνεια το θέμα, αλλά και η δικαιοσύνη ή το δικαίωμα των ίδιων θεσμικών οργάνων στο απόρριτο. Είναι σημαντικό λοιπόν οι πληροφορίες στην Ευρώπη να είναι κωδικοποιημένες και να είναι σταθερό στην προσέγγιση του εδώ διαμεσολαβητή. Στι κάτω χώρε το ίδιο έχω δει. Είναι χαρακτηρισμένε οι πληροφορίε εμπιστευτικέ και απόρριτε και για τον υπόλοιπο τη ζωή μα ξέρουμε ότι δεν θα δημοσιοποιηθούν ποτέ. Δεν είναι σωστό αυτό σήμερα με τι ε, ανάγκε που έχουν διαμορφωθεί. Είναι σημαντικό αυτό να αλλάξει. Και να έρθω και στο ερώτημα του κ. Βαλέσα που με, ευγενικά μου μετέφερε ο κ. Γιάρ Υπήρξε μια σημαντική υπόθεση στις κάτω ε, και για τους ε, αστυνομικούς, οι οποίοι ουσιαστικά ήταν θύματα των ε, προσταμένων τους και κυρίως θύματα διοικητικής συμπεριφοράς. Υπήρξαν κάποιες λαϊκίστικες ιδέες για το έργο τους στις κατοχώρες και υπήρξε ένας επικίνδυνος συνδυασμός και αρκετά λανθασμένος. Εγώ ήρθα σε επαφή με τον πρέσβη της Πολωνίας για το θέμα αυτό, για τους Πολωνούς εργαζομένους στις κάτω χώρες, το συζητήσαμε και κάποιες υποθέσεις έφτασαν στο γραφείο του Δημοσολαβητή. Από την άλλη, ένας πολιτικός ηθήνων θίξει το θέμα στις εφημερίδες ή στο κοινοβούλιο για τη διακριτική συμπεριφορά, θα μπορούσα επιτέλους και εγώ διεξιμοσολαβητής να τοποθετηθώ, να πω ότι δεν μ' αρέσει, ότι δεν το θεωρώ δίκαιο. Αλλά υπάρχει και ένα όριο. Διότι δεν μπορώ να περάσω σε πολιτική συζήτηση. Ίσως μία ή δύο φορές μπορώ να εκφραστώ με μεγάλη πυγμή, αλλά μετά θα πρέπει να σιωπήσω, διότι δεν είμαι πολιτικός. Και πρέπει να είμαι ιδιαίτερος προσεκτικός σε αυτό το τομέα. Ελπίζω να απήντησε ικανοποιητικά στο ερώτημα του κ. Βαλέσσα. Πρόεδρος, βεβαίως. Κύριε Μπρένιμπαγκερ, έχουμε ολοκληρώσει την ε, φάση της παρέμβασης των ε, μελών. Εάν θέλετε να προσθέσετε κάτι για να ολοκληρώσουμε, ε, έχετε το χρόνο. Ιδάλλως μπορούμε να κλείσουμε εδώ την ακροασή σας. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε. Ολοκληρώθηκε η πρώτη ακρόαση. Έχουμε τον δεύτερο υποψηφίο, τον κύριο Γέγκερ. Και με χαρά σας υποδεχόμαστε κύριε Γέγκερ. Σας ευχαριστούμε που υποβάλλατε την υποψηφιότητά σας. Θα γνωρίζετε ότι έχετε αρκετό χρόνο για την εισαγωγική σας ομιλία και μετά θα συνεχίσουμε με το χρόνο ερωτήσεων εντό εισαγωγικών για τα μέλη. Σας δίνω το λόγο για 10, 15 λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι βουλευτές, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω τα σημαντικότερα σημεία της υποψηφιότητάς μου και το όραμα για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Επίσης, Παράδειγμα τις ευκαιρία να ευχαριστήσω τους ευρωβουλευτέ από πέντε πολιτικές ομάδες και δέκα χώρες που με στήριξαν με τις υπογραφές τους. Διασυνοριακή και διακομματική στήριξη είναι πάρα πολύ σημαντική για την αξιοπιστία του διαμεσολαβητή. Ποια είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της υποψηφιότητά μου. Θεωρώ πώ έχει τέσσερα. Πρώτον, είμαι πραγματικά ευτυχής Ευρωπαίος, Γερμανός υπήκος, ε, μεγάλωσα και σπούδασα στη Γερμανία, εκεί ζει η οικογένειά μου. Η αγάπη με έφερε στην Γαλλία, παντρεύτηκα μια Γαλλίδα αρχιτέκτονα, τώρα η πατρίδα μου είναι η Γαλλία. Τα παιδιά μας σπουδάσανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία και τις Ηνωμένε Πολιτείε οικογένειά μου λοιπόν εκμεταλλευτήκε πλήρως όπως βλέπετε την ελευθερία μετακίνησης και εγκατάστασης. Δεύτερον, είναι η δουλειά μου να υπερασπίζομαι τις ελευθερίες των άλλων ανθρώπων. Το 1989 πήγα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Μόλις είχε πέσει το τείχος του Βερολίνου και ήμουν στην Μέκα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Νέε δημοκρατίες ε, έγιναν ε, κράτη-μέλη και θεωρεί το, το Συμβούλιο της Ευρώπης ο προθάλαμος τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι όροι που υπήρχαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτο δικαίου και τη δημοκρατία ήταν προαπαιτούμενα για τη διεύρυνση αυτή και βοηθήσαμε τι χώρε αυτέ να επιτύχουν τι προδιαγραφέ που έπρεπε. Ε, είχα εμπλακεί με αρκετά το Στην Αλβανία δεν υπήρχε Υπουργείο Δικαιοσύνη. Πήγα και βοήθησα να στηθεί ένα Υπουργείο Δικαιοσύνη. Οι χώρε έπρεπε επίση να να συντάξουν το διοικητικό δίκαιο, να φτιάξουν διοικητικά δικαστήρια και μου ζητήθηκε να προετοιμάσω ένα εγχειρίδιο με όνομα «Η διοίκηση και εσείς». Σε 50 σελίδες συνοψίζει τις αρχές του διοικητικού δικαίου της Δυτικής Ευρώπης. Η διαφθορά ήταν σοβαρή ανησυχία. Το Συμβούλιο της Ευρώπης προετοίμασε συμβάσεις αστικού και ποινικού δικαίου για να καταπολεμηθεί η διαφθορά. Και εγώ υπηρέτησα στην διεθνή ομάδα που συνέταξε αυτές τις συμβάσεις. Πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν κάποια ζητήματα για το αν τα κράτη-μέλη, τα νέα κράτη-μέλη, ε, κλήρωναν τις υποχρεώσεις τους και ο Γενικός Γραμματέας χρειαζόταν μια εμπιστευτική έκθεση. Ήμουν μέλος και της ομάδας η οποία συνέταξε αυτή την έκθεση. Αυτή ήταν η πρώτη δεκαετία στην οποία εργάστηκα επί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μετά πήγα να εργαστώ στην Interpol ε, ως επικεφαλής του νομικού τμήματος και εκεί πέρα ήμουν την 11η Σεπτεμβρίου. Τρίτον, ο διαμεσολαβητής είναι η ειδικότητά μου θα έλεγα. Επιστρέφοντας στο Συμβούλιο της Ευρώπης ε, εργάστηκα υπό τον πρώτο Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τον κύριο Χίλ Ρόμπλες, ο οποίος πριν ήταν ε, διαμεσολαβητής στην Ισπανία και είχε σχέσεις ε, με τους πρώην ομολόγους του. Οπότε σχημάτισα ένα δίκτυο του το λεγόμενο, και έφερα σε επαφή 40 διαμεσολαβητές από την Πορτογαλία στη Ρωσία και από την Νορβηγία μέχρι την Κύπρο. Εκπαιδεύσαμε το προσωπικό των διαμεσολαβητών ε, σε περιπτώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο να ανταλλάσσει πληροφορίες ε, και βεβαίως ε, στην δημιουργία θεσμών. Η Ένωση Διαμεσολαβητών της Μεσογείου που συστάθηκε από τους δημοσιολογητές της Γαλλίας, της Ισπανίας και του Μαρόκου για να στηρίξει την νότια ακτή της ε, Μεσογείου ιδρύθηκε και αυτή με δική μου συνεισφορά. Βοήθησα επίσης τη σύσταση του Ρώσου Διαμεσολαβητή και βοήθησα στην σύνταξη νομοθεσίας σε πάνω από έξι χώρες. Και βεβαίως υπάρχει και η Ιταλία και το Μονακό που δεν έχουν ακόμα καρποφορήσει αυτές τις προσπάθειες. Θα ήθελα λοιπόν να πω το εξή. Έχω φτιάξει ένα όνομα στον τομέα αυτόν. Τέταρτον, η ανεξαρτησία μου είναι το σήμα κατά τεθέν, εάν θέλετε. Η ανεξαρτησία είναι κάτι το σχετικό. Εξαρτάται από εσά, κυρίε και κύριοι βουλευτέ, να ορίσετε τον βαθμό ανεξαρτησία που θέλετε να έχει ο διαμεσολαβητή. Στην περίπτωσή μου, ο βαθμό ανεξαρτησία θα έλεγα πω είναι ο βέλτιστο όσον αφορά και πολιτικά κόμματα ομάδες συμφερόντων και χώρες ως ε, υπάλληλο σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς ε, ε, έδωσα βεβαίως την ενενομισμένη διαβεβαίωση για το θέμα αυτό πριν από 20 χρόνια και αυτό τον κανόνα τηρώ εδώ και 20 χρόνια. Ποιο είναι το όραμά μου λοιπόν για τον Ευρωπαϊκό Διαμεσολαβητή. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μία ανησυχία. Ανησυχώ γιατί πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτε δεν είναι τόσο τυχεροί όσο εγώ. Είχαν ελπίδε από την Ευρώπη για μια καλή ζωή, αλλά η ζωή του είναι δύσκολη. Και στην απελπισία του κατηγορούν την Ευρώπη για το ότι δεν ε, τηρεί τα υπεσχημένα και είναι έτοιμοι να παρετηθούν από την Ευρώπη. Προσωπικά δεν θεωρώ πω λιγότερη Ευρώπη θα βελτιώσει την κατάστασή του αντιθέτω. αλλά μια ε, πιο ανθρώπινη Ευρώπη θα το επιτύχει αυτό. Ε, πιο ανθρώπινη Ευρώπη σημαίνει πιο κοντά στους πολίτες της και τους κατοίκους της, θα τους αντιμετωπίζει με σεβασμό, θα ακούει τις ιδέες, τις ελπίδες, τις απαιτήσει τους και τα παραπονά τους. Η Ευρώπη η οποία δεν θα δίνει την εντύπωση πως κυβερνάται από πάνω προς τα κάτω και δεν έχει χώρο για πρωτοβουλίες. Τι μπορεί να κάνει λοιπόν ο μεσολαβητής. Υπάρχουν κάποιες ιδέες στις οποίες συμφωνούν όλοι, αλλά με διαφορετική χρειά θα έλεγα κάθε φορά. Και υπάρχουν προτάσεις που κάποιοι άλλοι δεν κάνουν. Η αποτελεσματικότητα πρώτα απ' όλα αντιμετώπιση των καταγγελιών. Η επίλυση ε, καταγγελιών δωρεάν, γρήγορα και με τρόπο δίκαιο δημιουργεί εμπιστοσύνη. Η συνεχής βελτίωση της αποτελεσματικότητας ε, της ε, δυνατότητας επίλυσης διαφορών επίσης ε, είναι ένας προφανής στόχος. Τώρα δεν θα αναφερθώ στον καταλογό των πιθανών μέτρων. Η σημασία επίση τη πρόληψη. Συμφωνούμε πω ο διαμεσολαβητή θα πρέπει να βοηθά τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συμπεριφέρονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε οι πολίτε δεν θα έχουν λόγο να παραπονούνται. Και αυτό, όπω επεσήμανε και ο κύριο ε, Διαμαντούρο, είναι μια διαδικασία χωρί τέλο. Και πάλι δεν θα επεκταθώ στα μέτρα, ε, αλλά θα ήθελα να επισημάνω πως οπωσδήποτε ο διαμεσολαβητής θα πρέπει να δώσει πρώτος το καλό παράδειγμα και να τονίσω τη σημασία των ερευνών που θα ξεκινούν με πρωτοβουλία του διαμεσολαβητή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τα ζητήματα των ουσιαστικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Επίσης η προληπτική συμμετοχή του διαμεσολαβητή στη δημόσια διαβούλευση που ξεκινάει η Κομισιόν θα εξαλείψει τις ε, αιτίες δημιουργίας καταγγελιών. Η δημοσιότητα. Η δημοσιότητα είναι που εγώ βλέπω τα πράγματα διαφορετικά σε σχέση με τους συνυποψηφίους μου. Η δική τους ανησυχία είναι η δημοσιότητα του διαμεσολαβητή. Όπως ε, σωστά επισημάνθηκε, αν δεν ξέρω κόσμος ότι υπάρχει ο διαμεσολαβητής δεν θα το χρησιμοποιήσει. Και διαβάζουμε με ενδιαφέρον για τους διάφορους τρόπους που προτείνονται. Κάποιους ομολογώ ότι δεν τους είχα καν σκεφτεί και ευχαρίστως να τους υιοθετήσω. Αλλά διαφέρω σε ένα βασικό ζήτημα η δημοσιότητα του διαμεσολαβητή δεν είναι ο αυτός σκοπός, είναι ένα μέσο. Ο πραγματικός στόχος είναι η δημοσιότητα ενός συστήματος. Ενός συστήματος που είναι δίκαιο και λειτουργεί σε γενικές γραμμές σωστά. Ένα σύστημα το οποίο έχει δικλίδες ασφαλείας, ένα σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει και θα ε, καθησυχάζει την κοινή γνώμη. Όπως είπε ο κύριος Φανρόμπαϊ στον κύριο Διαμαντερό. Εσείς κυρίε και κύριοι βουλευτέ είστε μέρος αυτού του συστήματος. Γι' αυτό η έμφαση που θέλω να δώσω εγώ είναι στη συνεργασία με εσά. Είναι στο, στη δημοσιότητα την δική σας. Γι' αυτό και οι προτάσει μου για να σας ε, παρέχω άμεσες αναλύσεις και πληροφορίες για καταγγελίες που προέρχονται από την χώρα σας ή την περιφέρειά σας ή αφορούν το τομέα που σας απασχολεί. Και έτσι θα επιμείνω σε καμπάνιες σχεδιασμένες ε, και που θα διεξάγονται με εσάς και τις εθνικές αντιπροσωπείες σας στις χώρες σας. Γι' αυτό προτείνω να στείλουμε προσωπικό από τις χώρες σας. αιτήματα για στήριξη, προτάσεις, ιδέες ε, κτλ. Γι' αυτό προτείνω να υπάρξει ένα σύστημα για να λαμβάνουμε αιτήματα για στήριξη, για προτάσεις, ε, ιδέες και λοιπές απαιτήσεις. Αυτή είναι μια ιδέα που δεν βλέπω να υιοθετούν οι συνυποψήφοι μου. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πως μπορούν να κάνουν όχι μόνο καταγγελίες, αλλά και, διάφορες, ε, και διάφορα αιτήματα να θέσουν στον νέο συλλογητή. Ο διαμεσολαβητής λοιπόν θα διοχετεύει τα αιτήματα αυτά στο αρμόδιο θεσμικό όργανο και εσείς και ο διαμεσολαβητής θα λαμβάνετε μια ε, ενημέρωση και ένα αντίγραφο για την συγκεκριμένη και λογική απάντηση. Και θα έχετε τη δυνατότητα να διαβιβάσετε τα αιτήματα αυτά εκεί όπου απευθύνονται. Και έτσι νομίζω θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την απογοήτευση των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και εδώ πέρα νομίζω πως ε, διαφέρω από τους συναδέλφους μου, είναι αφενός ε, το να βοηθάσουμε τις διοικήσεις των μελλοντικών κρατών μελών να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της προετοιμασίας των μεσολευτών και από την άλλη το θέμα είναι να γίνει γνωστή η λειτουργία της Διοίκησης Ένωσης πέρα από την Ένωση. Κάτι το οποίο τελικά δεν είναι και τόσο άσχημο για την ε, διακυβέρνηση 500 εκατομμυρίων ανθρώπων και βεβαίω συνεχώς βελτιώνεται. Αυτές είναι οι προτάσεις μου κύριε Πρόεδρε κύριε και κύριοι βουλευτές για την νέα φάση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Βασίζομαι λοιπόν στον κύριο Σέντερμαν, τον πρωτοπόρο και τον κύριο Διαμαντούρο, ο οποίο πραγματικά οικοδόμησε το θεσμικό αυτό όργανο, όπω σωστά τα είπε η κυρία Όμεν η προσωπική μου ανεξαρτησία, εμπειρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, συγκριτική γνώση θεσμικών οργάνων και η διεθνή μου εμπειρία νομίζω πω με καθιστούν ιδανικό υποψήφιο για αυτή τη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Thank you, Mr. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιάγκερ. Θα προχωρήσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Το λόγο έχει ο κύριος Γιάρ για το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Γιόγκερ. Καλώς ήρθατε στην ακρόαση. Γιατί εμείς, δηλαδή η Επιτροπή των Αφορών, είμαστε στο πλευρό του διαμεσολαβητή και οι δύο έχουμε στόχο να εξυπηρετούμε τον πολίτη. Οπότε να πω τη γενική μου παρατηρήση, θεωρώ πως και τα δύο θεσμικά όργανα είναι πάρα πολύ σημαντικά γιατί πάρα πολλοί πολίτες απευθύνονται σε εμάς ε, για την Ευρώπη. Οπότε το τι κάνουμε εμείς, αν το κάνουμε καλά ή όχι, έχει, ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αυτό αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Γι' αυτό καλό είναι που κάνουμε αυτή την ακρόαση. Το πρώτο ερώτημα αφορά την ανεξαρτησία, για ακριβώς γιατί παίζει τόσο σημαντικό ρόλο για εμάς για το τι σημαίνει ανεξαρτησία, πώς το ορίζουμε. Ήδη είπατε την άποψή σας, το ερώτημά μου είναι υπάρχει κάποιο όριο για εσάς. Υπό ερώτημα. Άκουσα πως κάποια κράτη-μέλη στο θέμα του διαμεσολαβητή ε, θεωρούν πως ο διαμεσολαβητής πρέπει να είναι ταυτόχρονα και βουλευτής να έχει μια λεγόμενη ουδέτερη έδρα. Ε, αυτό το θεωρείτε καλό ή όχι. Δεύτερο ερώτημα για το θέμα για το πρόγραμμα μάλλον για το ρώτησα και σε προηγούμενο στον προηγούμενο υποψήφιο ε, αν γίνεται ε, εμισολαπτής ποια είναι τα τρία σημαντικότερα πράγματα που θα κάνετε επόμενο ζήτημα Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Οπωσδήποτε σας απασχόλησε. Περιέχει πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας αφορούν και εμάς ε, στην Επιτροπή Αναφορών και πάρα πολλά ζητήματα αγγίζουν τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αλλά υπάρχει βεβαίως και το ζήτημα πως ε, λαμβάνουμε την απάντηση από την Κομισιόν πως ε, η χάρτα αυτή ισχύει όταν αφορά συγκεκριμένο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν είναι ικανοποιητική αυτή η απάντηση για εμάς. Εμείς θεωρούμε πως δεν γίνεται κάτι ουσιαστικό. Από την άλλη, από νομική σκοπιά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Τι άποψη έχετε για την αντίφαση και τελευταίο ερώτημα. Πώς θα βλέπατε τη σχέση μεταξύ Μεσολαβητού και Επιτροπής Αναφορών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε υποψήφι, κύριε Γέγκερ, είναι μεγάλη μου χαρά να σας ε, ακούσω σήμερα, ως υποψήφιου, δύο ερωτήσεις. Ως προς την ε, θεωρητική πλευρά του θέματος. Πρώτον, πώς ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής μπορεί να αποφασίσει και να εφαρμόσει ένα σαφή ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων. Αυτό είναι κάτι που επηρεάζει σοβαρά, όχι μόνο τη διαφάνεια και την καλή διακυβέρνηση, αλλά επιτρέπει να φτάσει κανείς και σε ψηλά επίπεδα διαφθοράς η απουσία του ορισμού. Αυτό είναι κάτι που να οριστεί και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και δεύτερον, εάν εκλεγείτε πώς ο μελλοντικός δημοσιολαβητής Γέγκερ θα δράσει σε περιπτώσεις παρόμοιες με το σκάνδαλο Πρίσμ. Ε, πώς ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής ο κύριος Γέγκερ, θα αντιμετωπίσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν περάσει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ για τη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών και απελευθέρωση του εμπορίου. Αυτό δεν είναι μια συνηθισμένη διαδικασία, αλλά φύγει ευαίσθητα προβλήματα όπω τα ανθρωπίνα δικαιώματα, η διαφάνεια, ε, ο ιδιωτικό βίο, η εμπιστευτικότητα και ευρωπαϊκού κανόνε που ορίζουν με σαφήνεια τι είναι δημόσιο και τι όχι. Και πώ οι, οι απόρριτε πληροφορίε μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από ποιον. Είναι απαραίτητο να οριστεί μια σαφής διαχωριστική γραμμή μεταξύ δημόσιων και απόλυτων πληροφοριών. Ειδικά στο σημερινό κόσμο όπου βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες εμπιστευτικές πληροφορίες να διαραίουν. Πληροφορίες που επηρεάζουν τον καθημερινό βίο των 500 ε, εκατομμυρίων πολιτών όπως είπατε κι εσείς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας. No, uh, uh, Ευχαριστώ κυρία Ματσόνη. Presentation. Ευχαριστώ τον ε, υποψήφιο που ήρθε να μας μιλήσει. Νομίζω ότι συμφωνούμε. Η σύγκρουση συμφερόντων αλλά και η ανεξαρτησία είναι στοιχεία τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά στο διοικητικό δίκαιο. Επομένως δεν είναι θέμα ορισμού. Ούτε συνδέεται το θέμα του ορισμού με το εσείς αν συγκεντρώνεται αυτά τα πρόσοντα έτσι για να είμαστε σαφείς τώρα. Εσείς Είστε έμπειρος, έχετε επιτελέσει σημαντικό έργο μέχρι τώρα. Αλλά για πέστε μας. Πώς βλέπετε τη λειτουργία αυτή, το λειτουργήμα τέλο πάντων. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις που καλείστε να πάρετε. Θα διαλέγεστε με πολύ σημαντικά θεσμικά όργανα θα κάνετε εχθρούς, ούτε μπορείτε να κάνετε πίσω. Θα πρέπει να δώσετε τη μάχη. Υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα προς τούτο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι προτάσεις σας. Κανείς δεν είχε τόσο ενδιαφέρουσες προτάσεις. Θα πρέπει να ακούτε όλους τους πολίτες. Έχετε προσπαθήσει όμως αυτό να το κάνετε. Να, αφού γκράζετε όλους, να απαντάτε σε όλους. Είναι υπέροχο αυτό, αν μπορείτε ένα τέτοιο σύστημα το εφαρμόσετε. Μακάρι, μακάρι, θα ήταν υπέροχο ένα τέτοιο σύστημα ακούσου. E. Κύριε Πάσκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ο κύριος Πάσκα. Κύριε Γέγκερ, έρχομαι και ρωτώ. Συνεργασία με τους εθνικούς διαμεσολαβητές. Εκπροσωπείτε τους πολίτες, όπως και θεσμικά όργανα, όπως και εκείνοι, και βέβαια το πνεύμα που θα το έργο σας θα παρομοιάζει με εκείνο των εθνικών διαμεσολαβητών. Άρα πώς θα συνεργαστείτε εάν εκλεγείτε με εκείνους. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τσίτσεστερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Γέγερ. Καλώς ορίσατε στην επιτροπή μας. Τονίσατε στην εισήγησή σας το θέμα της ανεξαρτησίας, της ουδετερότητας όπως πρέπει για έναν διαμεσολαβητή. Θα πρέπει όμως να πούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις το έργο του διαμεσολαβητή χαρακτηρίζεται από πολιτικοποίηση. Ιδίω εάν πρέπει να αναμετρηθείτε με κάποια αρχή εθνική ή ευρωπαϊκή για να υπερψηφίσετε πολίτη ή πολίτες. Οπότε, δεδομένου είπατε ότι είσαστε ένας ευτυχής Ευρωπαίος και λοιπά και λοιπά και φιλοευρωπαίος και όλα αυτά. Α, αυτό. Πώς θα λειτουργήσει στην περίπτωση που πρέπει να υπερευστείτε έναν απλό πολίτη. Γιατί θα πρέπει να μετρηθείτε με το κατεστημένο. Μία ερώτηση αυτή, δεύτερη ερώτηση. Αναγνωρίζετε τη δυσφορία που επικρατεί σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, εν μέσω πολλών Ευρωπαίων. Σίγουρα ισχύει μια τέτοια δυσφορία στον Ηνωμένο Βασίλειο που προέρχομαι. Και θεωρούμε ότι ό,τι ισχύει επειδή δεν δουλεύει τέλεια, δεν σημαίνει θέλουμε περισσότερη Ευρώπη, θέλουμε λιγότερη. Τέλος πάντων, Περισσότερη Ευρώπη σημαίνει περισσότερε καταγγελίε, περισσότερα προβλήματα μεταξύ πολιτών και αρχών. Άρα περισσότερη Ευρώπη, όπω είπατε, τι θα πει αυτό. Είναι κατά κάποιο τρόπο τέχνοντα για να εξασφαλίσετε περισσότερε αρμοδιότητε, περισσότερη δουλειά. Τρίτη ερώτηση. Τι θεωρείτε ότι είναι το πιο σημαντικό όπω έχετε πετύχει ή τέλο πάντων αυτό που σα συναντηπάζει περισσότερο. Πρόεδρος. Αυτή ήταν η τελευταία παρέμβαση και τον πρώτο γύρο τραπέζι, Οπότε σα δίνουμε τον λόγο να απαντήσετε στις ερωτήσει και κατόπιν πάμε στο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Γεια. για το ζήτημα της ανεξαρτησίας και τα όρια της. Μιλάμε για την ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή. Το σκέφτηκα αν ναι, έπρεπε να, να το πω αυτό που θέλω να πω ή όχι. Νομίζω πως μπορούμε να πούμε πως ε, ο νόμος ο οποίος ρυθμίζει αυτή τη στιγμή το θεσμικό όργανο του διαμεσολαβητή λέει μόνο πως θα πρέπει να έχετε στις υψηλότερες προδιαγραφές ε, ανεξαρτησίας. Και υπάρχει ένας όρκος και ορκίζεται ο δημοσιολαβητής ότι θα είναι ανεξάρτητος. Αλλά δεν ορίζεται το πώς. Δεν ορίζεται το τι θα γίνει ε, εάν υπάρχει ας πούμε καταγγελία εναντίον ε, ενός μέλους οικογένειάς του. Δεν ε, αναφέρεται το εάν πρέπει να, μπορεί να είναι μέλος κόμματος ή όχι. Δεν αναφέρονται τέτοια πράγματα και δεν θα σας τα πω εγώ. Εσείς πρέπει να ορίσετε πόση ανεξαρτησία θα δώσετε στον ε, διαμεσολαβητή. Έχω άποψη ξεκάθαρη, αλλά ο καθένας πρέπει να μείνει εντός των ορίων του. Ενδιαφέρον αυτό που είπατε για μια ουδέτερη έδρα στο Κοινοβούλιο. Κανένα πρόβλημα. Μια ουδέτερη έδρα είναι ουδέτερη έδρα. Ε, είναι κάποιος αυτομάτως ε, και άμεσα στη διεύθυνση του Κοινοβουλίου και αν είναι πραγματικά ανεξάρτητος ως παρατηρητής ε, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα από τις αρχές. Τα τρία σημαντικότερα ζητήματα τώρα του προγραμματός μου, οι τρεις προτεραιότητες. Το ένα είναι αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Μπρένινγκ Μάιρ, ότι θα πρέπει να μάθουμε την κατάσταση. Δεύτερον, επειδή ο χρόνος πιέζει, είναι το θέμα της δημοσιότητας και της άμεσης εμπλοκής στο πλευρό του Κοινοβουλίου και να παίξει ο διαμεσολαβητής τον ρόλο του. Και δεχτεί τον ρόλο και να μην προσπαθεί να ξεπεράσει. δεύτερη προτεραιότητα είναι η ανάλυση των περιπτώσεων και όταν γίνει η ανάλυση να δούμε αν υπάρχουν κάποια μοτίβα που σημαίνει πως υπάρχουν κάποιες προτεραιότητες. Τρίτη προτεραιότητα με συγχωρείτε, δεν μου έρχονται τα γερμανικά γιατί έχω χρόνια, δουλεύω χρόνια σε αγγλικά. Η τρίτη προτεραιότητα είναι να μην αφήνουμε τα μέλη μόνο τους. υπάρχουν ε, νομίζω πάρα πολύ μεγάλη δυνατότητα το προσωπικό να εξηγήσει στους πολίτες, ειδικά τη σημερινή εποχή, το ποιε είναι οι αξίες και το πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μου επιτρέπετε τώρα στα αγγλικά. Είπατε πώς σας προβληματίζει το γεγονός ε, πως όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, συχνά ο Διαμεσολαβητής και η Επιτροπή Αναφορών δεν μπορούν να κάνουν τίποτα λόγω της αρχής της επικουρικότητας. Ε, αυτοί είναι οι κανόνες. Τουλάχιστον εκεί όπου μπορείτε θα πρέπει να παραπέμπετε. Και βεβαίως αυτό δεν ισχύει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν ε, πολλά ουσιαστικά ανθρώπινα δικαιώματα στα οποία δεν έχει κάνει τίποτα αυτή τη στιγμή ο Διαμεσολαβητής εστιάζεται στα διαδικαστικά και όχι στα ουσιαστικά, αλλά μην ξεχνάμε πως ε, όσο αυτό είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να κάνουμε είναι να συνεργαστούμε με τα εθνικά θεσμικά όργανα και ειδικά τους διαμεσολαβητές για να φροντίσουμε τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων να γίνονται σεβαστά. Η σχέση μας τώρα με την Επιτροπή Αναφορών είναι ακριβώς το ίδιο πνεύμα. Ό,τι δεν μπορείτε να κάνετε εσείς πρέπει να το κάνουν διαμεσολαβητές και αντιστρόφως. Και αν δεν μπορούμε να το κάνουμε ε, πρέπει γρήγορα να παραπέμπετε στον Εθνικό Διαμεσολαβητή. Κύριε Μποσινάρου, πώς θα ορίσουμε τη σύγκρουση συμφερόντων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Νομίζω εδώ θίγεται δύο ζητήματα. Πρώτα απ' όλα τι πραγματικέ συγκρούσει συμφερόντων που μπορούν να αποδειχθούν και μετά το πώ αντιλαμβάνεται κανεί τη σύγκρουση συμφερόντων ή τον κίνδυνο, την απειλή σύγκρουση συμφερόντων. Το να αποδειχθεί αυτό είναι κάπω ε, δύσκολο. Αλλά το σημαντικότερο είναι ο κίνδυνο, δηλαδή η απειλή και η αντίληψη περί σύγκρουση συμφερόντων. Εδώ κάποιε φορέ έχουμε θέμα με, την, με το πώς θίγονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Λόγου χάρη, ο σύζυγος ή τα παιδιά σας ή οι εξαγχιστές συγγενείς σας μπορεί να εργάζονται σε ένα μέρος που είναι θύματα διακριτικής συμπεριφοράς. Εκεί πρέπει να ελέγξουμε το πώς η δική σας η οι ξανχιστε συγγενεις σας μπορει να εργαζονται περί ανεξαρτησίας ε, σχετίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα κατά την προσβολή τους. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα που θα πρέπει να το δει κανείς και να ορίσει και τα σχετικά όρια, ακόμη και για μέλη της οικογένειάς του. Για το σκάνδαλο πρίσμ. τι θα συνιστούσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει στι διαπραγματεύσει τη για τι ελεύθερε συναλλαγέ με τι ΗΠΑ. Με συγχωρείτε, αλλά έχω πολύ σαφεί προσωπικέ απόψει για το σκάνδαλο Prism. Και για μένα το πρόβλημα εδώ είναι τα διπλά μέτρα και σταθμά. Υπό πολλέ έννοιε. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί αντιλαμβάνονται κάποιον, τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ως υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που όμως από συγκεκριμένε συνθήκες είναι υπεύθυνο για αδίκημα που έχει σχέση με τα μέσα μαζική ενημέρωση και την ενημέρωση. Δεν θέλω να περάσω τώρα σε περισσότερε εξηγήσει, αλλά νομίζω ότι διπλά μέτρα και σταθμά είναι κάτι που είναι μια διαρκή απειλή. Η χρήση των απόρριτων πληροφοριών από άλλε χώρε. Υπάρχει εδώ ένα και μόνο κανόνα στο μυαλό μου. Ευρωπαϊκά πρότυπα πρέπει να εφαρμόζονται εδώ. Ακόμη και αν υπάρχουν υπερισχύοντες οικονομικοί λόγοι, θα πρέπει να μην ε, άρεται η προστασία. Είχε, υπήρχε και άλλο ένα ερώτημα για τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ ιδιωτικών και απόρριτων πληροφοριών, τα προσωπικά δεδομένα δηλαδή, και την προστασία τους. Εδώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε πολύ αυστηροί. Και πάλι έχουμε δύο μέτρα και σταθμά. Διαφάνεια από τη μια, προστασία από την άλλη και προστασία των, προσωπικών δεδομένων κυρίω. Εάν ε, γίνουν πολύ ελαστικά τα όρια τη προστασία προσωπικών δεδομένων, πάβει διαφάνεια, πάβει υπευθυνότητα που οφείλεται σε σχέση με τα θέματα αυτά. Ο Επίτροπο τη Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων πρέπει να το καλύπτει αυτό κατά την άποψή μου. Ο Ευρωπαίο Δημοσιολαβητή παραμένει ένα ενεργό μέρος στην λήψη σχετικών αποφάσεων. Κύριε Άουγκεν, σύγκρουση συμφερόντων και πω ορίζεται σε έναν ενδεχόμενο κώδικα καλής ε, διοικητικής συμπεριφοράς. Έχετε δίκιο εδώ. Εάν υπήρχε ένας τέτοιος κοινό κώδικας διαγωγής για τα θεσμικά όργανα και ήταν αρκετά συγκεκριμένο θα είχαμε λύσει εν μέρει το πρόβλημα. Πρέπει να πω όμω ότι κάπω επιφυλάσσουμε ω προ αυτή τη βεβαιότητα. Διότι όπω όλου του νόμου, όσο πιο πολύ συγκεκριμένο είναι κανεί, τόσο πιο πολύ δυσκολεύεται να καλύψει κάτι που δεν το είχε συλλάβει, σκεφτεί, δεν το είχε περάσει από το νου όταν ε, συνέτασε τον νόμο. Μπορεί να προκύψουν λοιπόν περιπτώσεις για πράγματα που δεν τα έχουμε σκεφτεί. Και εκεί επειδή θα ε, είναι εκτός του πεδίου όσων καλύπτει ο νόμος, ε, θα υπάρχει δυσκολία. Για το ρόλο του δημοσιολαβητή, λόγου χάρη. Υπάρχει αυτό το, αυτή η νομική ασάφεια, λόγου χάρη, με την προσχώρηση και την ε, συνδρομή σε πολιτικά κόμματα. Τη στήριξη από πολιτικά κόμματα. Οπότε είμαι υπέρ ενός κώδικα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει στο τέλος να υπάρχει μια τέτοια διατύπωση που να παραμένει ανοιχτή σε πολλές ερμηνείες για να επιτρέπει να καλύπτονται και πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Πράγματα που δεν έχουν καλυφθεί ήδη, δεν τα έχουμε σκεφτεί ως σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει στη σύγκρουση συμφερόντων, όπως είπα, να λαμβάνουμε όπως στην περίπτωση και την ε, απειλή καθώς και την αντίληψη. Θέλατε ένα παράδειγμα για σκληρές αποφάσεις που έχει λάβει ο διαμεσολαβητής χρειάστηκε να λάβω μια πολύ δύσκολη απόφαση όταν ήμουν επικεφαλής της νομικής υπηρεσίας της Ιντερπολ. Κάποιος, πολύ γνωστός, ήταν ιδιοκτήτης ρωσικού καναλιού. Ε, συμμετείχε στον, ε, ενεχόταν στον πόλεμο κατά της Τσενίας και υπήρχαν κατηγορίες στη Ρωσία αναντίον του για, για κατάχρηση για διαφθορά, ό,τι θέλετε. Οι αρχέ τη Interpol ζήτησαν λοιπόν ένταλμα για τον άνθρωπο αυτό έπρεπε να αποφασίσω αν είναι πολιτικό, πολιτική δίωξη ή επί της ουσίας, πραγματική. Αποφάσισα ότι είναι πολιτική η δίωξη, ειναι πολιτικη διωξη παρολο που δεν μπορούσα να αποκλείσω ότι υπήρχαν και οικονομικοί λόγοι και μάλιστα βάσιμοι. Ζήτησα λοιπόν να μην συλληφθεί ο άνθρωπος αυτός, το ζήτησα και από τον Γενικό Γραμματέα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορούσε το δικό μου πεδίο αρμοδοτήτων. Ήταν όμω πάρα πολύ δύσκολη απόφαση, πολύ σκληρή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να αρνηθώ αυτή την απέτηση μια μεγάλη προσωπικότητα που ερχόταν από τη ρωσική πλευρά. Είπατε κι εσεί είναι πολύ δύσκολο να αφήνει κανεί να ξεφεύγουν οι διάδικοι του. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ρεαλιστικό να καλύπτονται τα αιτήματα όλων των πολιτών που θέτουν ερωτήσει. Εγώ όμω έχω μιλήσει με αρκετού ευρωβουλευτέ και το έχω ήδη σχολιάσει. Ε, κάποιοι έχουν έναν εκατομμύριο ψηφοφόρου. Και βλέπουν ότι δεν μπορούν να συζητήσουν με όλου, δεν μπορούν να καλύψουν όλε τι αιτήσει που φτάνουν σε αυτού. Πιστεύω λοιπόν ότι ο διαμεσολαβητή θα πρέπει να παίχει κάποιε φορέ, να μην δέχεται όλα τα αιτήματα και να προσπαθήσει να βρει και έναν τρόπο να διοχετεύει τα αιτήματα αυτά στου αρμόδιου. Δεν μπορεί κανεί να είναι τέλειο, δεν μπορεί να καλύψει τα πάντα. Μπορεί όμω να ομαδοποιεί υποθέσει οι οποίε μπορούν να ε, απευθύνονται στη συνέχεια στι αρμόδιες αρχέ. Άλλωστε, για να μπορεί κανεί να ασχοληθεί με προσφυγές πρέπει να ξέρει ποιο κάνει τι. Ο διαμεσολαβητή ακριβώ όπω την κατεύθυνση πρέπει να εργάζεται, όχι να αφήνει του ευρωβουλευτέ μόνο του και να εξυπηρετεί του Ευρωπαίου πολίτε, ε, βοηθώντα του να αποταθούν στο σωστό άνθρωπο. Κύριε Πάσκα, για τη συνεργασία με του εθνικού διαμεσολαβητέ. Είναι απλό. Υπάρχει ένα δίκτυο Ευρωπαίων Δημοσιολαβητών. Ο κύριος Διαμαντούρος το ίδρυσε. Υπάρχουν αξιωματικοί σύνδεσμοι εδώ και υπάρχει πολύ, δυνατότητα, πολύ γρήγορη δυνατότητα διασύνδεση με τηλεφωνή μετά με ε, ηλεκτρονική αλληλογραφία. Όλα τα κανάλια είναι ανοιχτά. Και υπάρχει μια ελαφρά διαφορά σε σχέση με το έργο του Δημοσιολαβητή. Και μια μικρή δυσκολία ότι γι' αυτό χρειάζεται συγκατάθεση του πολίτου που έχει αποταθεί σε σας. Εδώ πρέπει να είναι κανείς πολύ προσεκτικός. Αλλά μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις άλλες πλευρές, τις εθνικές, τους εθνικούς διαμεσολαβητές, για τη διαδικασία, για την απόκριση. Για το, ε, εάν θα ενημερωνόμαστε για το πώς επιλήθηκε η υπόθεση. Εδώ, ω Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής, αλλά και εσείς ως Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να ξέρω εάν οι υποθέσεις αυτές έχουν τελικά επιληθεί μέσω του δικτύου εθνικών δημοσιολαβητών ή εάν εν τέλει ο πολίτη που σας είχε αρχικά αποταθεί δεν έλαβε καμία απάντηση μετά από όλες τις προσπαθίε του. Και Τσίτσεστερ. Ανεξαρτησία. Για πόσο χρόνο και σε τι βαθμό θα μπορούσα να είμαι ανεξάρτητος εάν κάτι συμβεί που έχει πλήρως πολιτικό χαρακτήρα. Αυτό συνδυάζεται με όσα είπε προηγουμένως για τη δημοσιοδίκηση. Πιστεύω ότι θα ήμουν ανεξάρτητος. Αυτό ελπίζω. Και προσωπικώς, αν αναλάβω αυτή τη θητεία, και επειδή θα κρατήσει μόνο ένα χρόνο η θητεία μου μέχρι να λήξει και η δική σας, εάν επανεκλεγώ και τεθεί θέμα ανεξαρτησίας, εάν κάποιος ε, έχει τέτοιο θέμα, θα πρέπει πριν το τέλος της θητεία του να παρατηθεί. Δεν πρέπει να τηθεί καν τέτοιο θέμα για τον ευρωσκεπτικισμό σε όλε τι ευρωπαϊκέ χώρε και τη δική σα που λέει ότι χρειαζόμαστε λιγότερη Ευρώπη. Και τι πιστεύετε εσείς ότι μπορώ να κάνω εγώ ως υπόθεση εργασία για να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη στο έργο μου. Το περισσότερο... Ναι, ναι, ναι, από την άποψη των δεδομένων υπάρχει δυνατότητα αύξησης περισσότερη δουλειά για το διαμεσολαβητή, εντάξει, αλλά ταυτόχρονα κάτι που λειτουργεί καλά. Δεν έχει να κάνει με το πόσε πολλέ προσφυγέ επιλύει κανεί. Οπότε δεν είναι θέμα μεγέθου η καλή διοργάνωση, αλλά καλή οργάνωση. Η καλύτερη διοίκηση βεβαίω και θα οδηγήσει σε μείωση των προσφυγών και το αντίστροφο για τα μεγαλύτερα μα επιτεύγματα δεν έχουν σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώ. Είναι πολύ πρόσφατα. Το 2008, βάσει νόμου, 750 πολίτε τη Ρωσική Ομοσπονδία έλαβαν το δικαίωμα να κάνουν κάτι που ποτέ δεν του είχε επιτραπεί. Να πάνε σε κέντρα, σε σοφρονιστικά ιδρύματα και να δουν τι συμπεριφορά έχουν εκεί οι υπόδικοι. Πώς τους μεταχειρίζονται τους φυλακισμένους. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό, γιατί χρειάστηκε μεγάλη συνεργασία με τις ρωσικές αρχές, ώστε και η Γερμανία και οι κατοχώρες και η Δανία και το Ρωσικό Εμπορικό Επιμελητήριο να μου δώσουν τα απαραίτητα κονδύλια για να εκπαιδευτούν αυτοί οι 750 άνθρωποι. Και μάλιστα να μην υπάρξουν δυσκολίε με τι αρχέ. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο. Είναι ένα επίτευγμα για το οποίο είμαι ιδιαίτερα περήφανο. Ιδιαίτερα για τη χώρα μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιάνγκερ για το δεύτερο γύρο. Πρώτο. Η κυρία Κολάρας Καπουμπίνσκα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η εμπειρία σας. Συμβουλή της Ευρώπης κλπ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και κυρίως έτσι Βλέπουμε το θέμα σε πολλές ευρωπαϊκές γωνίες, πολύ ενδιαφέρον. Το βασικό έργο του Δημοσιολαβήτη είναι τα προβλήματα του κόσμου, επίση ε, το να συνεργάζεται με θεσμικά όργανα που τα πηγαίνει σε αυτό το μέτωπο πολύ καλά και ο Διαμαντούλος. Επίσης, στην εισήγησή σας τονίσατε το έργο του Διαμεσολαβητή όσον αφορά τις ε, γειτονιάζουσες, τις υποψήφιες για ένταξη χώρας. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Συνεργασία δηλαδή με διαμεσολαβητέ, όχι μόνο με χώρες μέλη, αλλά και με τις γειτονιάζουσες χώρες. Με τις οποίες έχουμε προγράμματα συνεργασίας, έχουμε την γειτονική πολιτική, την πολιτική προσανατολάς κλπ rule of law and citizens issues are very much neglected. So... Uh, και επομένω, επί τη βάση όλων αυτών, θα κάνουμε την επιλογή μα, γιατί πάντω ε, αυτή τη δραστηριότητα του Δημοσιολογητή είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά τώρα έχω και μία ερώτηση. Μα αναφέρατε ότι η ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή είναι κάτι το οποίο δεν διέπεται από κάποια ρύθμιση. Και τελικά είναι θέμα εμείς πόσο θέλουμε να τον απελευθερώσουμε, του λύσουμε τα χέρια, αλλά ακριβώς ε, κάποιος που βγάλει αποφάσεις θα πρέπει να παράσχει την ανεξαρτησία σε κάποιο τέτοιο θεσμικό όργανο. Άλλωστε, ο νομοθέτης μπορεί να μεταβάλει άποψη. Σας ρωτώ επομένως, μήπως χρειάζεται να ε, υποστεί νομοθετική ρύθμιση το ζήτημα της ανεξαρτησίας του διαμεσολαβητού, μια που τώρα δεν υπόκειται σε τέτοια ρύθμιση από την Αμερία. Βέβαια, ε, η υπερβολική νομοθετική ρύθμιση δεν είναι τόσο καλή, αλλά ε, νομίζω ότι κύριε πρόεδρε συγχαρητήρια κύριε Γέγκερ εξαιρετική η θα είναι κάτι το θετικό. Κάσμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια κύριε Γέγκερ. Εξαιρετική η εισήγησή σας. Έχουμε συναντηθεί και η δουλειά σας για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι παράδειγμα προς μίμηση. Πάντως, όπως είπαν και οι θα πρέπει να τα δούμε ελαφρά διαφορετικά, από κάπως διαφορετική οπτική γωνία. Έχετε δίκιο. Υπάρχει κάποια αποστασιοποίηση των ε, Ευρωπαίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οπότε και νομίζω ότι εάν διαμεσολαβητή βάλουμε κάποιον πρώην διαμεσολαβητή, τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα όσον αφορά αυτό το πρόβλημα. Πάντω τώρα συγκεκριμένα, για να δούμε το θέμα εκείνο το οποίο απασχολεί εμένα και το μισό κοινοβούλιο όσον αφορά την, την, την, την προσβασιμότητα σε έγγραφο πλαστού κοινού, τη διαφάνεια κλπ. Πώ θα γίνει αυτό, δεν θα πρέπει να πετύχουμε την σωστή ισορροπία, σωστή ισορροπία μεταξύ αφενό αποτελεσματική λήψη αποφάσεων πλευρά μικρών οργάνων και από την άλλη μεριά το δικαίωμα των πολιτών να γνωρίζουν πώς διαμορφώνται αυτές οι αποφάσεις. Και κατά τον τρόπο να μπορούν να αποδοθούν ευθύνε ή στα θεσμικά όργανα. Ε, ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Μπούλαμ. σας ευχαριστώ. Αλλά στην συνέλευση ΑΚΕ είχα κάποια υποχρέωση, την Ευρωπαϊκή να μιλήσω. Ξέρω τη διαδρομή σας, έχουμε ήδη συναντηθεί. Έχω μόνο μία ερώτηση να σας θέσω. Πέραν αυτών που ρώτησαν οι συνάδελφοι. Πέστε μας, σε σχέση με το δίκτυο των διαμεσολαβητών, με απασχολεί αυτό πάρα πολύ. Γιατί νομίζω ότι έτσι έχει την ευκαιρία ο κάθε Ευρωπαίος, παντού σε όλη την Ευρώπη, και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Το πρόβλημα είναι ότι δύο από τι 27 χώρε δεν έχουν διαμεσολαβητή. Εσεί τι μπορείτε να κάνετε. Αυτό το ερώτημα προκύπτει συνέχεια σε σχέση με εμένα. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε πλήρη κάλυψη, πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ισότητα, δηλαδή να μπορούν όλοι οι Ευρωπαίοι να μπορούν να διαμαρτυρηθούν, να, να καταγγείλουν κάποιες αποφάσεις που δεν τους έχουν σεβαστεί. Επίσης, τι θα γίνει με την ανισότητα στον ρόλο των ε, διαμεσολαβητών. Ας πούμε στη Γαλλία δεν είναι δυνατόν να προσφύγει κανείς κατά κάποιας κρίσης ε, αποφάσεις, κάτι το οποίο αλλού στην Ευρώπη δεν ισχύει. Δεν ξέρω και, και ο Ευρωπαίος Δημοσιοπτής δεν μας το Πόσο μας μπορεί να μια τέτοιου είδους εναρμόνιση για αυτή την πλευρά των δραστηριοτήτων. Επομένως και ποιοτικά και γεωγραφικά. Τι μπορούμε να κάνουμε. Ο ε, Μπουλό ήταν ο τελευταίος που έλαβε το λόγο. Οπότε σας ξαναδίνουμε την ε, σκητάλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κυρία Κουλάσκα Μπομπίνσκα. Θέλω το εξής να σας πω. Θεωρήσατε πάρα πολύ θετικό το ότι έχω συνεργαστεί με θεσμικά όργανα εκτός των μελών, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και κάτι το οποίο δεν θέλω να το ακούω συχνά. Δηλαδή τα προβλήματα με τα θεμελιώδη δικαιώματα στις χώρες αυτές που προαναφέραμε. Στη Σερβία και αλλού έχουμε διαμεσολαβητέ που έχουν ε, ισχυρή προσωπικότητα και ε, ευξημένες αρμοδιότητε και οι οποίοι μπορούν να σηκώσουν το κεφάλι τους από την άλλη μεριά όμω. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα. Δεν θέλατε να πείτε αυτό. Αλλά το ακούω συχνά. Εμεί προωθούμε τα ανθρώπινα δικαιώματα εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά. Όμω στο περιβόλι μας δεν προσέχουν το τι γίνεται. Ε, αυτό εγκυμονεί κινδύνους. Τώρα, ο λόγος που θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι κάνουμε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σημαντικό. Έχουμε την εξωτερικές δράσεις και εσείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορείτε να απαιτήσετε για τον σεβασμό των δικαιωμάτων. Όμως, για να είμαστε αξιόπιστοι, θα πρέπει οι χώρες αυτές, τις οποίες πιέζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και θέλουν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει ανά πάσα στιγμή, λέγω, να πείσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Διοίκηση είναι δίκαιη έχει διαφάνεια κλπ. Επομένω, συμφωνώ 100% μαζί σας. Άλλη ερώτηση ήταν το κατά πόσον θα πρέπει να έχουμε κάποιο είδου ε, νομοθετική ρύθμιση, χωρίς παραθυράκια, ε, ξεκάθαρη για την ανεξαρτησία του διαμεσολαβητή. Δεν μπορώ παρά να πω ναι σε μια τέτοια πρόταση. Έχω εδώ πέρα σχετική τεκμηρίωση. Ας πούμε αν έχουμε κάποιο συγγενή, κάποιο δημοσιολογητή ο οποίος ε, εργάζεται σε κάποιο θεσμικό όργανο ε, το οποίο ερευνά ο τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Ιδίω αν είναι στο νομικό τμήμα ή σχετικό ο συγγενής. Ε, τότε ο δημοσιολογητής θα πρέπει να δηλώσει το τι συμβαίνει. Από την άλλη μεριά, ε, αν δεν κάνει τίποτα δεν ρωτήσει, αυτό δεν είναι καλό για τον πολίτη. Ε, Επομένω θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, ε, πλήρης και ξεκάθαρη νομοθετική ρύθμιση για την εξαρτησία. Κύριε Κάσμα, ευχαριστώ για τα καλά σα λόγια. Και εγώ να σα πω ότι θα πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και μεταξύ ε, απόδοσης ευθυνών και λογοδοσία. Τώρα, η λήψη αποφάσεων προϋποθέτει αυτό το οποίο είπαμε, κάποιο, την σφαίρα του ιδιωτικού βίου σε σχέση με το θεσμικό όργανο. Εάν κάποιοι συνεργάτες δεν μπορούν να συζητήσουν, δεν μπορούν να εκφραστούν, δεν μπορούν να πούν κάτι το οποίο να μην καταγράφεται κάπου συνέχεια, ε, τότε ε, πάμε προς κάποιο είδους στήρα διαδικασία λήψη αποφάσεων, γιατί τότε δεν έχουν καλή στάθμη στον υπέρ και τον κατά. Δηλαδή, εάν όλα γίνουν σαν τόσα συζητούνται η λήψη απόφαση, τότε θα έχουμε κάποιο δυσφορία από πλευρά ε, του κόσμου. Ναι, χρειάζεται πλήρη ε, διαφάνεια. Αλλά από ένα σημείο και μετά αυτό επηρεάζει την αποτελεσματική αποφάσεων. Επομένω, μέχρι πού θα πρέπει να φτάσουμε σε αυτό το μέτωπο. Γιατί έρχεται κάποια στιγμή κατά την οποία η διαδικασία λήψη αποφάσεων είναι Ιωνία, άτυπη. Σε σχέση με το τι ισχύει σήμερα ποτέ και αν έχουμε την εσωτερική εμπλοκή των όσων παρτίζουν τον μηχανισμό λήψη αποφάσεων, αυτό αν κάποια στιγμή δημιουργηθεί πλήρω και αν αποκτήσουν προσβασιμότητα οι πολίτε, αυτό είναι καλό. Αλλά όμω αυτό δεν θα πρέπει να γίνεται ευθύ εξ αρχή τη διαδρομή. Αυτό αφορά κάθε διοίκηση. Επομένω θα πρέπει ο μεσολαβητή να, να ξέρει σε ποιο σημείο τη διαδρομή θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο. Αλλά θετικό αυτό που ρωτήσατε. Αυτό όμω βέβαια έχει να κάνει και με το είδο του εγγράφου. Ένα email. Τα email μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο πρόσβαση. Ότι όμω σημειώνεται σε ένα χαρτάκι, ε όχι, αυτό δεν αποτελεί αντικείμενο πρόσβαση. Επομένω έχουμε κάποιου κατόφλι ε, τήρηση κάποιων τύπων πριν από το οποίο ή μετά από το οποίο κάτι δημοσιοποιείται ή αντίστοιχα δεν δημοσιοποιείται. Κύριε το δίκτυο των δημοσιολογητών έχει κάποια κενά. Τα κενά είναι κάποιες χώρες που δεν έχουν δημοσιολογητή. Κάπου υπάρχει Επιτροπή Αναφορών, στην άλλη χώρα που το ξέρω τι έχει. Και πολύ ορθώς είπατε ότι από πλευρά του πολίτη σε αυτές τις χώρες δεν υπάρχει ενδικό μέσο, δεν υπάρχει μέσο τέλο πάντων προσφυγής κατά δικαστικών αποφάσεων. Τι κάνουμε. Ο διαμεσολαβητής προσφύγεται τα δικαιώματα. Όχι κάποια δικαιώματα, εν γέννη τα δικαιώματα. Γιατί το λέω αυτό, διότι υπάρχουν κάποιε συμφωνίες, συμβάσεις, οδηγίε κανονισμοί που ορίζουν τη συγκρότηση ανεξαρτήτων οργάνων των διοικητικών αρχών, ούτως ώστε να ρυθμίζεται το τι γίνεται Φερρυπίν σε μια περίπτωση δεσμή διάκριση σε κάποια χώρα. Και επομένω, ήταν τον αυτό να γίνει. Για τον ισολογητή. Δεν το αποκλείω. Και επίση έχετε δίκιο ότι αυτή τη στιγμή η εντολή αυτών των διαμεσολαβητών διαφέρει πάρα πολύ από χώρα σε χώρα. Άρα θα πρέπει πρώτα πρώτα να συμφωνήσουμε τι θέλουμε να διέπει τους διαμεσολαβητές και κατόπιν θα πρέπει να επιβάλλουμε το να ισχύσουν αυτά. Δεν νομίζω ότι αυτό μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Γιατί τα νομικά συστήματα διαφέρουν πάρα πολύ, νομικές παραδόσεις διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός 200 ετών. Είναι αναπόσπαστο τμήμα αυτού του δικαϊκού συστήματος και στη Γαλλία επίσης συνάντησε μεγάλα εμπόδια η θέσπιση αυτής της θέσης και μόλις τώρα άρχισε σιγά σιγά να προσαρμόζεται η Γαλλία. Επομένω, αυτό το οποίο είπατε θα γίνει, αλλά όχι σύντομα. Θα πρέπει να πιστούν οι χώρες ότι θα πρέπει να μπορούν να πειράσουν το, τα πράγματα οι δημοσιογραφητές όπως έγινε με, τον κύριο Διαμοντούρη και την Τουρκία γιατί προσπαθούσε επί μεγάλο διάστημα ο κύριος Διαμοντούρος να πείσει την Τουρκία να έχει διαμεσολαβητή. Και νομίζω ότι έγινε την πλάστηκα η προσπαθή του Διαμαντούρ στο να προσχωρήσουν σε, αυτό, σε αυτή την πρόταση. Στο να έχουν τέλο πάντων οι Τούρκοι. Έχει κάποιο όριο η προσπάθεια αυτή που κάνουμε για την ε, εναρμόνιση τη ρύθμιση. Και όσον αφορά επίση τι διαφορέ των ομοδιότητα των διαμεσολαβητών, εδώ ας εμπιστευτούμε εκείνους, διότι εκείνοι έχουν υπόψη τους τις ε, αρμοδιότητες των συναδέλφων τους γύρω γύρω και οπότε έχουν επομένως αυτό ως επιχείρημα έναντι των αρχών της χώρας τους. Κάπως αυτό και για τη Γαλλία. Ο Δημοσιολογητής είχε κάπως ε, λιγότερες αρμοδιότητες από ό,τι άλλους στην Ευρώπη. Ε, τώρα επομένως ε, αναβαθμίστηκε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε κύριε Γιέγκερ. Δεν θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος να λάβει το λόγο, οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ την ακρόασή σας. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Έχετε πέντε ακόμη λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κατά πρώτον θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τα γερμανικά μου. Έπειτα ολοκληρώνοντας τη συζήτηση. Κάθομαι και σκέφτομαι τι έμαθα εδώ. Διότι ήρθα με τις δικές μου απόψεις εδώ και τελικά ήρθα αντιμετώπως με τις δικές σας ιδέες και απόψεις. Όταν λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να επανακαθορίσω τις αυτοτεραιότητές μου, αυτό θα παίξει μεγάλο ρόλο. Νομίζω ότι η διαχωριστική γραμμή μεταξύ του τι είναι πολιτικού χαρακτήρα και τι όχι είναι κάτι που θα πρέπει να το ξανασκεφτώ πολύ σοβαρά. Ο δημοσιολαβητής θα πρέπει να μένει τελείως αμέτωχος ε, υποθέσεις που υπάρχει και μια ελαφρά οσμή πολιτικής απόφασης ε, θα πρέπει να το ξανασκεφτώ και αυτό και δεν βρίσκω ότι θα είναι τελικά εποφελές. Δεν πρέπει να είναι τόσο ντροπαλός ο Μεσολαβητής, ούτε να κρύβεται πίσω από τη, τα επίσημα όρια της θητείας του. Θα πρέπει να διακινδυνεύει και κάποια πράγματα ε, ενώπιν των άλλων θεσμικών οργάνων και λίγο να πιέσει. Να πιέσει την όλη προσπάθεια ε, άσκησης των αρμοδιοτήτων του. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα σημαντικό παράδειγμα που με αφορά άμεσα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο γύρο προτάσεων της Τρόικας για την Κύπρο. Δεν υπήρχε περιθώριο ένας δημοσιολαβητής να επισημάνει, να επισημάνει, όχι να αποφασίσει, να επισημάνει το ενδεχόμενο ότι μπορεί να παραβιάζονται εδώ θεμελιώδη δικαιώματα πολιτών και ενδεχομένω να επηρεάσει τη λήψη μιας τέτοια απόφαση. Θα έπρεπε να πει ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητής ότι η Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει να μην φτάσει κανείς σε προχωρημένη ηλικία σε συνθήκες ένδυας. Κάποιοι μπορεί να είχαν αποταμιεύσει στις τράπεζες εκεί που θα γινόταν η, η ανάληψη των θα έπρεπε λοιπόν να το επισημάνει. Το ενδεχόμενο ότι κάποιος μπορεί ακόμη και να εξετάζει την ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων κάποιων εντό εισαγωγικών πολιτικών αποφάσεων, το πώς αντίκεινται αυτές τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι σημαντικό. Θα συμφωνήσω τελικά μαζί σας. Ο Ευρωπαίος Δημοσιολαβητή έχει φωνή και έχει μια φωνή που θα πρέπει να ακούγεται περισσότερο στα ζητήματα ανθρωπίνων των δικαιωμάτων παρά να ασχολείται μόνο με θέματα καλή διοίκηση, διοικητικά ζητήματα πρόσβαση σε πληροφορίε και λογοδοσία πρέπει ε, να εκδίδει συστάσει που είναι δεσμευτικέ για όλου, για όλα τα θεσμικά όργανα και θα πρέπει να λέει κάποια πράγματα επί τη ουσία και ε, με μεγάλη σαφήνεια. Νομίζω λοιπόν ο διαμεσολαβητή είναι αυτό που θα πρέπει να ασχολείται με τέτοιε υποθέσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γέγκερ. Χειροκροτήματα. Καλή σα τύχη. Colleagues, we have συνεχίζεται η συζήτηση. Καλώς ορίζει την κυρία Όμαν Ράιτεν. Και... Την ευχαριστώ για την παρουσία της θα έχει εκείνη το λόγο για 10 με 15 λεπτά για να μας παρουσιάσει την υποψηφιότητά της. Και μετά θα περάσουμε στις ερωτήσεις και θα δώσουμε τον λόγο στους βουλευτές. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Γιατί είναι, είναι ακόμα επίσημη γλώσσα. Έτσι, και αν μιλούσα αγγλικά, 430 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν έχουν τα αγγλικά ως πρώτη γλώσσα. Λοιπόν, Έχω απαντήσει τις ερωτήσεις, τώρα η ακρόση αυτή μου δίνει την ευκαιρία να πω λίγα πράγματα για το άτομό μου, την εμπειρία μου και τα προσόντα που θεωρώ πως με καθιστούν ε, κατάλληλοι για το αξίωμα αυτό. Βεβαίως, αναμένεται να πω και κάτι για το πώς βλέπω εγώ τη μελλοντική λειτουργία του διαμεσολαβητή. Λέω του διαμεσολαβητή, αλλά είναι και τρεις γυναίκες βεβαίως ε, υποψήφιες. Ο λόγος, ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους είμαι υποψήφια είναι η ιδιαίτερη εμπειρία που είχα την ε, επίλυση διαφορών. Μέχρι τον Ιανουάριο ήμουν πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών στην Ολλανδία. Ο οργανισμός αυτός που ξεκίνησε το 1985 ήταν πάρα πολύ μικρός αρχικά τότε και επεκτάθηκε υπό προεδρίας μου και αυτή τη στιγμή υπάρχουν 54 τέτοιες επιτροπές επίλυσης διαφορών που καλύπτουν ένα ολόκληρο φάσμα ασχολούμαστε και με την διαμεσολάβηση και με δεσμευτικές γνωμοδοτήσεις και μπορώ με υπερηφάνεια να πω πως ο οργανισμός αυτός στην Ολλανδία ήταν και υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την εναλλακτική επίλυση διαφορών. Νομοθετήσαμε για τον ΟΝΤΙΡ και ΑΝΤΙΡ, δηλαδή εναλλακτική επίλυση διαφορών και επίλυση διαφορών στο διαδίκτυο και ο οργανισμός μας ήταν ε, παρόν και σε πολλές ε, ε, επισκέψεις και ακροάσεις. Και η εμπειρία που είχα εκεί νομίζω πως μπορώ να τη χρησιμοποιήσω και στην δουλειά μου ως δημοσιολογητής. θα να σας πω λίγα πράγματα για εμένα. Από το 1981 είμαι βουλευτής, τα πρώτα 8 χρόνια, με τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και μετά ε, από το 89 και μετά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, οπωσδήποτε έχω μια δική μου ομάδα, οι άνθρωποι που ε, θα δουλέψουν ε, μαζί μου νομίζω είναι γνωστοί από τους διάφορες υποθέσεις που έχουμε χειριστεί. Η αφετηρία μου είναι και τώρα κάθε μέρα πώς πρέπει να σκεφτόμαστε, να έχουμε κατανόηση για κάθε άποψη, σεβασμό για κάθε άποψη και έτσι να ε, σχηματιστούν γέφυρες για να υπάρχει η κατάλληλη πολιτική επιπλέον. Πάνω απ' όλα προσανατολίζουμε στα αποτελέσματα. Και, όπως και εσείς που είστε αίρετοι, έτσι και εγώ θέλω το καλύτερο αποτέλεσμα για τους πολίτες. Το προσωπικό μου σύνθημα στην πολιτική ήταν πάντα διαθέσιμη, κοντά στον πολίτη και αυτό προκύπτει από ένα δικαίωμα δικαιοσύνης και ε, βεβαίως ε, από ένα αίσθημα αγάπης για τον άνθρωπο. Γιατί λοιπόν είναι σημαντικό το αξίωμα του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή. Θεωρώ πως πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερο βάρος στην εμπιστοσύνη του πολίτη προς την ευρωπαϊκή πολιτική. Γιατί οι πολίτες αντιμετωπίζουν αποφάσεις που λαμβάνονται στην Ευρώπη και έχουν συνέπειες στην καθημερινή τους ζωή. Για τη δουλειά τους, ε, για τη σύνταξή τους, ε, και βεβαίως ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής ε, δεν ε, λύνει τα προβλήματα, αλλά το θεσμικό αυτό όργανο μπορεί να βοηθήσει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, γιατί ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει πως υπάρχει κάποιος ο οποίος βοηθάει, ο οποίος ακούει, πως έχει στραμμένο το αυτί του και διορθώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάει συγνώμη εκεί όπου αυτό απαιτείται. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής λοιπόν βοηθάει στην αλλαγή της κουλτούρας της διοίκησης. Γιατί θα πρέπει η διοίκηση να είναι ανοιχτή, να έχει διαφάνεια, να λαμβάνει τις σωστές ε, αποφάσεις και να επιδεικνύει υπευθυνότητα και να δίνει τις πληροφορίες, να παραδέχεται τα λάθη, θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη προς την εξυπηρέτηση από πάνω, από την κορυφή μέχρι τα κατώτατα κλιμάκια. Από το Ευρωβαρόμετρο του 2011 φαίνεται πως οι πολίτες εκτιμούν ιδιαίτερα την ορθή διοίκηση και τις καταγγελίες που μπορούν να κάνουν. Και το άρθρο 297 της συνθήκης λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια διοίκηση ανοιχτή και ανεξάρτητη. Και θεωρώ πως, όπως λέει και το Ευρωβαρόμετρο, 42% των Ευρωπαίων πολιτών θεωρούν πως είναι αρκετά ανοιχτή η διοίκηση. Άρα ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι αυτός ο οποίος θα βοηθήσει τους πολίτες να βρουν το δίκαιο τους. είναι ο συνήγορος πολίτη. Πραγματικά ζούμε τώρα πώς λειτουργεί ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Τα τελευταία χρόνια έχει νομίζω γίνει ένας ε, σημαντικός εταίρος του Ευρωπαίου πολιτικού. ο κύριος Σέντερμαν και ο κύριος Διαμαντούρος έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και πάνω εκεί θέλω να βασιστώ κι εγώ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα μείνουμε σε αυτά. Όχι, θα αφιερώσω την ενέργεια και τη δημιουργικότητά μου έτσι ώστε η βάση αυτή, η σωστή, να επεκταθεί και θεωρώ πως αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη συνεργασία και την εμπλοκή του Κοινοβουλίου. Και θα έλεγα πως ε, θα βασιστώ στα εξής στοιχεία για την κράση. Πρώτα απ' όλα στην δημοσιότητα, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας αν δεν ξέρει ο πολίτης ότι υπάρχουμε ή αν δεν ξέρει ε, ποιες είναι οι αρμοδιότητες που έχεις. Και αν παραδείγματο χάρη την έκθεση του 2012 πως ε, είχαμε ε, γύρω στις ε, ε, καταγγελίες και 700 όσες από αυτές ήταν ε, εκτός της ε, εντολής θεωρώ πως έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη πρόκληση οπότε πρέπει βεβαίως να δούμε τι θα γίνει με το site κτλ αλλά νομίζω πως μπορούμε να καταβάλουμε ακόμα μεγαλύτερες προσπάθειες και άρα θα πρέπει ο διαμεσολαβητής να είναι γρήγορος και αποτελεσματικός γιατί όταν έρχεται με μια καταγγελία προς τον διαμεσολαβητή ο πολίτης θέλει μια γρήγορη απάντηση και διαπιστώνω πως ο χρόνος αντιμετώπισης καταγγελιών κατά μέσο όρο είναι 11 μήνες, αλλά σε ένα τρίτο των περιπτώσεων ε, διαρκεί πάνω από ένα χρόνο η διαχείριση των καταγγελιών. Οπότε εγώ θα καταβάλω μια προσπάθεια να μειώσουμε ακόμη περισσότερο τον χρόνο ε, απάντησης. Και θα προσπαθήσουμε, όπως είπα, να δίνουμε μία απάντηση. Δεν ξέρω αν θα επιτύχουμε τους τρεις μήνες, αλλά νομίζω πως μπορούμε να επιτύχουμε μία συμφωνία κυρίων για να είμαστε πιο γρήγοροι. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε, και είχα και την εμπειρία στην σχετική υπηρεσία στην Ολλανδία, ότι όταν ε, κάνει μια καταγγελία ένας πολίτης έχει ένα νούμερο φακέλου και κάθε βήμα στον φάκελο αυτόν μπορεί να μπαίνει σε ένα ψηφιακό σύστημα για να το βλέπει ο πολίτης για να έχει άμεσα τις πληροφορίες για την κίνηση της υπόθεσής του. Κυρίες και κύριοι, ένα τρίτο σημείο είναι το τι πρέπει να κάνει ο διαμεσολαβητής στο θέμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ε, κάτι το οποίο με απασχολεί. Γιατί η χάρτα αυτή ε, βρίσκεται στην ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας και πρέπει να ισχύει πλήρως και για τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τις αποκεντρωμένες υπηρεσίε και άρα θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η ευρωπαϊκή διοίκηση. Αυτά θα πρέπει να είναι στο DNA, να είναι καθημερινή υπόθεση των θεσμικών οργάνων. Ο διαμεσολαβητής παίζει έναν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το θέμα. Και όχι μόνο στα άρθρα 41 και 42, αλλά συνολικά επιπλέον και στο καταστατικό του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή αναφέρεται η συνεργασία με τα θεσμικά όργανα των κρατών μελών για να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών και όπως ε, είπα ξανά για το ευρωβαρόμετρο, φαίνεται πως 85% των Ευρωπαίων πολιτών έχουν ε, ελλειπή γνώση για το θέμα αυτό. Οπότε, εάν ε, γίνω διαμεσολαβητής, θα αφιερώσω πάρα πολύ ενέργεια σε αυτό το θέμα. Τέταρτον, η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Διαμεσολαβητού το Κοινοβούλιο και ειδικότερα η Επιτροπή Αναφορών και ο Ευρωπαίος Διαμεσολογητής είναι, κατά την άποψή μου, ε, φυσική σύμμαχη. Οι στενές επαφές με την Επιτροπή Αναφορών θεωρώ άρα πως έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία και όχι μόνο με την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης. Αλλά Εγώ είχα πει πως ε, σε 6,5 χρόνια είχαμε 18 ειδικέ εκθέσεις. Πρέπει να τον δούμε αυτόν τον αριθμό. Δεν σημαίνει αυτό πως πρέπει κάθε μήνα να έχουμε μία έκθεση, αλλά πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούμε τα μέσα που έχουμε στην ε, διάθεσή μας. Κατόπιν, κυρίες και κύριοι, ένα άλλο θέμα. Και αυτό είχε αναφερθεί και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκό Κώδικα Ορθής Διοικητική Συμπεριφοράς. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, καταλήξαμε σε συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή στον οδηγό αυτό ορθής διοικητική συμπεριφοράς. Και θυμάμαι και τη συνεργασία και με την κυρία Μαργκό Κέσλερ. Αυτό έγινε το 2001. Θεωρώ πως για όλα τα θεσμικά όργανα πρέπει να υπάρχει ένας τέτοιος οδηγός. Αυτό το οποίο δηλαδή πρέπει να έχουμε είναι, αν μου επιτρέπετε, ένας κανονισμός ευρωπαϊκού διοικητικού δικαίου. Γιατί αν έχει άλλο κώδικα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άλλο το κάθε θεσμικό όργανο, τότε δεν υπάρχει διαφάνεια. Θεωρώ πως η εμπειρία εδώ πέρα του διαμεσολαβητή ε, και το τι μπορεί να προσφέρει, ε, στο και αν δεν είναι εντός αυτής της θητείας, ε, είναι νομίζω το να καταλήξουμε σε μια διοργανική συμφωνία για αυτό το θέμα. Κυρία Πρόεδρε, αυτά ήταν τα ζητήματα τα οποία είχα εγώ να αναπτύξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ομενράιντεν. Και τώρα αρχίζουμε με τους συντονιστάς. Πρώτον, ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ κύρια Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Ομενρόιτεν. Έχω γράψει εδώ πέρα από αυτά τα οποία είπατε, το δέσμευση για να εργαστούμε για τους ανθρώπους για το τι πρέπει να κάνει ο διαμεσολαβητής ή η διαμεσολαβητής εν πάση περιπτώσει. Αυτό νομίζω πως είναι ξεκάθαρο και συμφωνούμε σε αυτό και εμείς ε, και η Επιτροπή Αναφορών. Και πραγματικά είχαμε σε αυτό τη δέσμευση όλων των υποψηφίων. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω το εξή. Τα τρία σημαντικότερα πράγματα που θα κάνετε αν αναλάβετε αυτό το αξίωμα, όπως ρώτησα και τους άλλους ε, συνυποψηφίους σας. Πού θα δώσετε έμφαση. Το άλλο θέμα βεβαίω αφορά τι δημοσιότητα πρέπει να δοθεί στον διαμεσολαβητή, το αναφέρατε. Πρέπει να υπάρχει ε, μεγαλύτερη δημοσιότητα. Εδώ πέρα συμφωνούμε και έχουμε και εμείς ένα παρόμοιο πρόβλημα σε Επιτροπή Αναφορών. Και ένα άλλο ερώτημα, πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη δημοσιότητα αυτή. Για τη χάρτα τώρα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ένα θέμα το οποίο βεβαίως μας απασχολεί συνεχώς και στην Επιτροπή μας και σωστά είπατε πώς έχουν τα πράγματα. Εμείς έχουμε το πρόβλημα πως ε, ε, καταγγελίες πηγαίνουν ε, στον διαμεσολαβητή. Κάτι το οποίο βέβαιω είναι αφενός δικαιολογημένο, αλλά από την άλλη η χάρτα μπορεί να εφαρμοστεί όταν περάσει στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάλι λοιπόν υπάρχει ένα έλλειμμα εδώ πέρα. Αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκό δίκαιο, διαπιστώνουμε συχνά πως είναι δίκαιο το αίτημα, η καταγγελία, η αναφορά, αλλά δεν έχουμε κάποιο νομικό μέσο για να κάνουμε κάτι. Τι θα κάνετε εσείς γι' αυτό το πρόβλημα χάρτα ανθρωπίνων πέντε δικαιωμάτων και μετά αρμοδιότητες στα κράτη-μέλη. Και τελευταίο ζήτημα συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών. Νομίζω αναφέρθηκε ήδη. Δεν χρειάζεται καν να το θέσω σε ερώτημα, αλλά θα ήθελα να ισχύσει όντως κάτι τέτοιο στην πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Ε, Γεια, ευχαριστούμε λέει Πρόεδρος. Ο κ. Κάσμαν για τους σοσιαλιστές. Κύριε Μοναράκη, συγχαρητήρια όσον αφορά την εισήγησή σας, τις οποίες άκουσα μόνο τα δύο τρίτα. Ε, θα ήθελα κάτι να σας πω πάντως όσον αφορά ε, το σχολείο κ. Μποστινέρο. Σωστό αυτό που να υπάρχει ε, γρήγορη απόκριση στα θέματα των πολιτών, οπότε αυτό, θα πρέπει να το αλλάξετε αν, λάβετε τα καθήκοντά σας και όσον αφορά τώρα το χάρτη των, δικαιωμάτων, ε, συμφωνώ, έχετε δίκιο, αυτό να ισχύει για όλα. Τα θεσμικά όργανα αυτό θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μα συνεχώ. Τώρα, με δεδομένο ότι αυτό ισχύει μόνο στο κοινωτικό δίκαιο α, άμεσα, Εσεί πώ θα μπορούσατε αυτό τον προβληματισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα να το εφαρμόσετε, να διαπνέει τι αποφάσει σα και να διαπνέει και τι σχέσει σα με τα θεσμικά όργανα. Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο αναφέρατε όσον αφορά αυτόν τον κώδικα διοικητικής διοντολογίας και επίσης ε, σωστά επενέσατε την ε, κυρία Κέστρε τη συνάδελφό μας που έχει επιτελέσει τόσο σημαντικό έργο. Επίσης έχετε δίκιο όταν είπατε ότι υπάρχει ε, φυσική συμμαχία μεταξύ Κοινοβουλίου και διαμεσολαβητού, ώστε πρέπει να υπηρετούμε του Ευρωπαίους. Επίσης τι γίνεται σε περίπτωση που υπάρχει μια σύγκρουση, αντίθεση, δηλαδή δεν συμφωνεί η Κοινοβουλία και η διαμεσολαβητή για κάποιο θέμα που αφορά του πολίτε. Εσεί τι προσέγγιση θα είχατε, κάτι άλλο τώρα σε σχέση με αυτό που ο κ. Μποσινάρ. Καλά, έχουμε πάρα πολλέ ερωτήσει, αλλά νομίζω ότι υπάρχει επικάλυψη μετά όσο είπε ο κ. Ε, Γιάρ. Εσεί τι θα συμβουλεύετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν, ε, για παράδειγμα, ε, είχαμε να διαμαντευτούμε μια εμπορική συμφωνία ας πούμε, με τη ΣΥΠΑ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λοιπόν και τον Άουκεν. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Εγώ θέλω να επισέλθω στην ουσία, σε κάτι που με προβληματίζει. Υποψήφοι δηλαδή που συνδέονται με απευθείας με κάποιο κόμμα. Νομίζω ότι είπατε στην εισήγησή σας ότι πόσο συνδέεται τέλο πάντων το ότι όλοι εκλεγήκαμε εδώ με κάποια πολιτική πλατφόρμα και εσείς το ίδιο. Το θέμα είναι κατά πόσον θα ακούσετε το τα αιτήματα αυτών που σας εξέλιξαν. Δεν ξέρω, μήπως δεν μεταφράστηκε σωστά από τα Ολλανδικά. ίσως έγινε μπέρδεμα στο πέρασμα του, του, του, του, κειμένου από τα Ολλανδικά στα Δανέζικα. Πάντως έχω εδώ πέρα κάτι άλλο το οποίο έχετε γράψει στην European Voice, το οποίο με εξέπληξε πρώτα-πρώτα. Εκεί μας λέτε ότι η ανεξαρτησία ενός δημοσιολαβητή είναι το ίδιο όπως η ανεξαρτησία ενός επιτρόπου. Όμω, όλοι ξέρουμε ότι είναι πολιτικό ο διορισμό ή ο ορισμό του επιτρόπου. Επί τη βάση και εθνικό συμβάρδενο ο διαμεσολαβητής θέλει, πρέπει να έχει μια ανεξαρτησία όπως ο δικαστής. Κάτι το οποίο είναι όλος διάφορο. Οπότε, όταν μας λέτε ότι η πιο σωστή για να γίνουν μεσολαβητέ, είναι κάποιε σαν και εμά. Νομίζω ότι μπερδεύεται το ρόλο του μεσολαβητή με τον ρόλο ενός πολιτικού. Οπότε, Εντάξει, ε, το να έχετε χρηματίσει ευρωβουλευτή και μετά να κάνετε ένα διάλειμμα και μετά να γίνετε δημοσιογραφητή δεν πειράζει. Αλλά έτσι κατευθείαν αφού διακηρύσετε ότι προσέχετε την εξαρτησία θα πρέπει και να είστε ανεξάρτητοι, να φαίνεστε ανεξάρτητοι. Ενώ εμείς εδώ εκπροσωπούμε πολιτικά κόμματα. Γι' αυτό και με εκπλήσει ο ορισμός της εξαρτησίας που δώσατε. Επίσης μας λέτε για αυτού του είδους την νομοθετική ρύθμιση, για την κώδικα διοντολογία κλπ. Για την διοίκηση. Έτσι βλέπετε την εξαρτησία. Όταν λέτε ότι η σύγκρουση των συμφερόντων δεν είναι αντικειμενική διαπίστωση. Κάτι γνώμη μου. Θα πρέπει να είναι αντικειμενική αξιολόγηση η σύγκρουση των συμφερόντων. Κάτι δηλαδή διαφορετικό από το, από το πώς λειτουργούμε εμείς εδώ. τόσο αφορά τη διαφάνεια. Βλέπω ότι είχατε απόσχε τις ψηφοφορίες το 1049 τότε που ψηφίσαμε. Άρα με εκπλήσει το πώς ε, θέλετε τώρα να γίνει η Μεσολαβήτρια και ενώ δεν στηρίξε το Κοινοβούλιο στην προσπάθειά του ε, για, τον, ε, για τον 1049. Επίσης όπως ρωτήσαμε για τον άλλο υποψήφιο, τι λέτε για, την συμφωνία, τη συνθήκη του, του Άρχους το αφορά περιβάλλον και θέλουν πολλοί να μπλακούν περισσότερο. Ε, Κάτι το οποίο στο 1049 ήδη προβλέπεται. Άρα, εσείς θα μπορέσετε να ενισχύσετε το ρόλο του πολίτη σε σχέση με ε, αυτές τις ρυθμίσεις. Και αν ναι, τότε γιατί είχατε απόσχεση στη σχετική ψηφορία. Ευχαριστούμε κυρία Βέρτμαν. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα. Ευχαριστώ. Να θέσω δύο ερωτήματα. Το πρώτο αφορά έναν... προέρχεται από συνάδελφο της ομάδας μου και το πρώτο από κυρία Όκεν περί διαφάνειας μπορείτε να αναπτύξετε το γιατί είχατε απόσχεση σε αυτό το τόσο σημαντικό θέμα της διαφάνειας και ποια είναι η άποψή σας για την αναθεωρήση του κανονισμού που αφορά την ε, πρόσβαση την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έπειτα στην παρουσίασή σας ενώπιν της ομάδας Άλντε, είχατε πει ότι θα είστε ανεξάρτητοι και ότι θα είστε μια υποψήφιο που θα το εξασφαλίσει αυτό. Πώ θα το συνδυάσετε αυτό με την ψήφο σα στην τότε ψηφοφορία για την υποψηφιότητά σα για Ευρωπαίο και Μεσολαβητή. Και ακόμη μια ερώτηση. Είχαμε πολύ δύσκολε δημοσιονομικέ συζητήσει και διπλωματεύσεις αυτή την περίοδο τη Ευρωπαϊκή κρίσης και τη Ευρωπαϊκή οικονομίας σε κρίση. Πώς βλέπετε το έργο σας σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουν προκύψει, διότι δημοσιολαβητής έχει ένα συγκεκριμένο κονδύλι στη διάθεσή του, δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτό το όριο, οπότε πώς θα κάνετε πιο αποτελεσματικό το έργο σας. Πώς θα βελτιώσετε την αποτελεσματικότητα από τη μια και από την άλλη, πώς θα επιτύχετε περισσότερα προς όφελος των Ευρωπαίων πολιτών. Πώς το βλέπετε αυτό, μπορείτε να μας δώσετε την ε, τοποθέτησή σας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Τσίτσος δεν είναι στην αίθουσα. Λοιπόν. Ίσως να κλείναμε τον πρώτο γύρο με τους συντονιστές και να ξαναδώσουμε το λόγο στην κυρία ε, Ομεν Ρότεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Βέτμαν, η πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα για μένα. Και ως διαμεσολαβητής πρέπει να αποδεχθώ το κανονισμό του Κοινοβουλίου. Ως υποψήφια δεν θέλω να επηρεαστώ από την συζήτηση που διεξάγεται. Ξέρω ότι υπάρχει και συζήτηση γιατί η πρόσβαση του κοινού είναι ένα θέμα. Η διαφάνεια είναι άλλο. Πώς όμως να παραμείνουμε και να τα συνδυάσουμε σε αυτό το θέμα και να τα συνδυάσουμε με τα προσωπικά δεδομένα. Αυτό είναι όλη η συζήτηση στο Κοινοβούλιο. Εκεί υπάρχει όλη η διαμάχη και ο διχασμός. Όμως, σε αυτήν τη φάση δεν φτάσουμε υπέρ κάποιες πλευράς. Ο διαμεσολαβητής δεν τάζεται υπέρ καμίας πλευράς. Είναι αρμόδιος και υπεύθυνο μόνο με, για τη χάρτα και όσα ορίζουν το 45 και το 42. Περί διαφάνειας και πρόσβασης του κοινού. Υπάρχουν εκκρεμείς αποφάσεις εδώ. Και επίσης ο διαμεσολαβητής για αυτά αποφασίζει. Για τις δημοσιονομικές ε, περικοπές και τους περιορισμούς. Νομίζω ότι μπορεί να είναι κανείς αποτελεσματικότερος σε σχέση με το τι γίνεται σήμερα και να είναι τόσο αποτελεσματικός όσο σήμερα. Από τη γνώση μου τώρα και από την εμπειρία μου στην Επιτροπή Αναφορών ξέρω ότι υπάρχουν πλέον και ψηφιακές δυνατότητες. Μπορεί λοιπόν να είναι κανείς αποτελεσματικότερος όσο ποτέ. Και νομίζω ότι θα ήταν συνετή ιδέα εάν κοιτάζαμε τον ιστότοπο του διαμεσολαβητή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Επιτροπής ε, Αναφορών, για να δει πόσο καλύτερη συνεργασία θα μπορούσαμε να έχουμε μεταξύ των δύο. Μπορούμε να διευκολύνουμε η μεν το έργο των δε. Βεβαίω λοιπόν υπάρχουν δημοσιονομικοί περιορισμοί, υπάρχει ένα κονδύλι, προβλέπεται ένα συγκεκριμένο ποσό, ούτε θα υπάρξει ποτέ αύξηση, αλλά ούτε θα συζητηθεί ποτέ κάτι τέτοιο από μένα, περισσότερα από όσα προβλέπονται τώρα. Κυρία Άουκεν. Κυρία Άουκεν, κάνατε πολλές παρατηρήσεις για την ανεξαρτησία. Αναφέρατε από την εισαγωγή μου κάποια πράγματα, αυτό λεξη και είναι και στα αγγλικά, θα σας τη στείλω, η παρατήρηση την οποία κάνατε Ε, υπάρχει εκεί πέρα. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι πως η ανεξαρτησία αποδεικνύεται τη στιγμή που κάποιος αναλαμβάνει ένα αξίωμα. Και αυτό βεβαίως αποδεικνύεται για, ε, και πρέπει να αποδειχθεί βεβαίως γιατί ορκίζεται και κανείς ενώπιον του 10 ότι θα είναι ανεξάρτητος. Στο δε κοινοβούλιο είχαμε συχνά την συζήτηση όσον αφορά το διορισμό του διαμεσολαβητή για το εάν θα πρέπει να έχει κάποια πολιτική σχέση με κάποιο πολιτικό χώρο και θα ήθελα να σας πω πως και ο κύριος Σέντερμαν και είναι πραγματικά τέλειο παράδειγμα, από τη στιγμή που ανέλαβε τα καθήκοντά του, δεν μας απασχόλησε ξανά το ζήτημα αυτό και μάλιστα τον επανεξελέξαμε. Και είχε βεβαίως κάποια σχέση με πολιτικό χώρο. Οπότε, κυρία Αουκέν, θα έλεγα πως η εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντική. Κοιτάξτε, αν δεν μπορώ να σας πείσω, εντάξει, στο κοινοβούλιο έχει ο καθένα την άποψή του εδώ πέρα και ψηφίζει όπως θέλει να ψηφίσει. Αλλά θα έλεγα πως μπορείτε να έχετε εμπιστοσύνη, μου, εμπιστοσύνη πως εάν εκλεγώ θα είμαι ανεξάρτητη. Οι υποψήφοι ε, εδώ πέρα που ήρθαν όλοι, ούτως ή άλλως, έχουν κάποιοι, ε, κάποια εξάρτηση από το κοινοβούλιο, γιατί από εσά θα εκλεγούν και ο καθένας από εσά θα πρέπει να ζυγίσει ποιον ψηφίζω και αυτόν τον οποίο ψηφίζω πρέπει να σκεφτώ πραγματικά μπορεί να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των πολιτών που εκπροσωπείτε εσείς ε, κύριε Κάσμαν, εσείς κύριε Μαρτίνες, εσείς κύριε Άουκεν. Αυτό πρέπει να κάνετε και ο διαμεσολαβητής δεν είναι πολιτικός και αυτή τη στιγμή γίνει διαμεσολαβητής δεν είναι πλέον πολιτικός και έχει τελείως διαφορετικές ε, ε, προτεραιότητες από αυτές τις οποίες πιθανώς είχε πριν. Ως διαμεσολαβητής είναι κανείς ανεξάρτητος, εκφύσεως Έτσι, και δεν απαιτείται πλέον. Όπως είπα, απαιτείται ένας τελείως διαφορετικός ρόλος και φροντίζει για να υπερασπίζει τα συμφέροντα των πολιτών. Κύριε Κάσμα τώρα, στα γρήγορα. Ναι, αλλαγές. Ναι. Συμφωνία κυρίων με τα θεσμικά όργανα για τις απαντήσεις. Θα το εξετάσω. Το είπα και στην ομιλία μου. Χάρτα. Η χάρτα. Η χάρτα δεν είναι κάτι που εγώ μόνο πρέπει να έχω στο νου μου. Όχι κάτι που πρέπει να είναι πάντοτε στο νου όλων μας, αλλά να βρίσκεται και στο γονότυπο όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Πρέπει να τους πείθω καθημερινά φυσικά ότι αυτό πρέπει να είναι μια διαρκής διαδικασία. Έπειτα Είπατε ότι υπάρχει φυσική συμμαχία μεταξύ τη Επιτροπή Αναφορών και του διαμεσολαβητού. Τι θα γίνει αν υπάρξει σύγκρουση μεταξύ των δύο όμω. Ελπίζω ένα από τα πρώτα θέματα που θα αναλάβω να είναι κάτι που και το Κοινοβούλιο θα το στηρίξει. Η απόδειξη της ανεξαρτησίας μου. Τέλος. Τοποθέτηση για την Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών. Ο διαμεσολαβητής. Δεν είναι νομοθέτης. Άρα, εσείς το κοινοβούλιο θα αποφασίσετε για το θέμα αυτό. Έτσι. Μπορεί να υπάρξει η πολιτική η ανθρώπινη, η διαμεσολαβητική αν θέλετε τοποθέτηση βάσει της χάρτας. Όμως δεν μπορεί να παρέμβει στην νομοθετική διαδικασία ο διαμεσολαβητής. Μην ε, να γι' αυτό. Κύριε Γιάρ. Αναφερθήκατε στο αξίωμα του διαμεσολαβητή. Μόνο στα γερμανικά νομίζω υπάρχει αυτή η λέξη που αναφέρατε. Ο συνήγορος του πολίτη. Μα εγώ πάντα έτσι αισθανόμουν. Και μπορώ να το αποδείξω κιόλα. Γιατί πάντα ε, εκλεγόμουν με τις δικές μου δυνάμεις. Και δεν εκλέγεται κανείς, ούτε και στην Ολλανδία, εάν δεν έχει κάποια σχέση με τους πολίτες. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για μένα αυτό το αξίωμα, γιατί θα ήθελα οι πολίτες, οι Ευρωπαίοι, που ασκούν τόση κριτική στην Ευρώπη, να έχουν την αίσθηση πως υπάρχει κάποιος που μας ακούει Υπάρχει κάποιος που διορθώνει τα θεσμικά όργανα και φροντίζει από τον Σιρορό μέχρι τον κύριο Μπαρόζο ή τον κύριο Φανόμποη όλοι να είναι προσανατολισμένοι στην εξυπηρέτηση του πολίτη. Αυτό πρέπει να, γνωρίζουμε. Και μετά ρωτάτε πώς σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. Ε, και να δώσω δημοσιότητα. Πρέπει να δούμε πώς και δεν είναι γνωστός ο διαμεσολαβητής στην Ευρώπη. Πώς και δεν γνωρίζουν το τι κάνει ακριβώς ο διαμεσολαβητής. Θεωρώ λοιπόν πως η επικοινωνία, τα ΜΜΕ, αλλά και η συνεργασία με την Επιτροπή Αναφορών είναι πάρα πολύ σημαντική. Θεωρώ, παραδείγματος χάρη, πως πρέπει να δούμε και το site. Γιατί υπάρχουν νέες δυνατότητες τώρα. Αν προσκαλέσω εγώ... Αν ε, φορτώσω ένα site, ε, περνάνε πάρα πολλά δευτερόλεπτα, ενώ θέλει 400 μιλισεκόντια για να φορτώσω το Google. Γλώσσες επίσης. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Αλλά θεωρώ πως μπορούν πολλά πράγματα να βελτιωθούν. Έχουν μπει οι βάσεις, τώρα πρέπει να ε, επεκτάθηκε από τον κύριο Διαμαντούρο, αλλά τώρα πρέπει να βελτιωθεί η επικοινωνία. Πώς θα γίνει αυτό. Με πυθό. Με μεσολάβηση. Και με μηνύματα. Να φροντίσουμε να υπάρξει μια σωστή λύση. Μια ανοιχτή συζήτηση, ένας ανοιχτός διάλογος, αλλά και αν δεν γίνει αυτό πρέπει να το λέμε. Και θα φροντίσω, εάν εκλεγώ, να μην εκπροσωπώ μόνο τους υπαλλήλους στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά να είμαι παρούσα εκεί πέρα, τακτικά, γιατί έτσι μπορεί κανείς να αντιληφθεί καλύτερα τα μηνύματα του κόσμου. Ευχαριστούμε. Να περάσουμε στο δεύτερο γύρο. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Μπουλόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητή Ρία, γνωριζόμαστε. Μία ερώτηση λοιπόν θα κάνω, που την έθεσα και στον προηγούμενο υποψήφιο. Δηλαδή, το δίκτυο των Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών. Δεν έχουν ακόμη όλα τα κράτη-μέλη Ευρωπαίοι μεσολαβητη ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες παρόμοιες δομές σε κάποια κράτη. Αυτές παρόλα αυτά δεν επιτρέπουν εθνικό διορισμό, ούτε εθνική εκπροσώπηση. Και είναι δύσκολο να έχουν τον ίδιο ρόλο τις οι ενδιάμεσες δομές όπως ένα διαμεσολαβητή. Η ερώτησή μου είναι η εξή. Νομίζετε ότι ο Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μπορεί να ασκήσει επίδραση, επιρροή σε αυτά τα κράτη-μέλη που δεν διαθέτουν ακόμη διαμεσολαβητή, ώστε να προβλέψουν κάτι ανάλογο. Και αυτά τα κράτη που δεν έχουν σήμερα και τα μελλοντικά. Πιστεύετε ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να φροντίσει να αναλάβουν τις απαραίτητες αρμοδιότητες οι διαμεσολαβητές σε εθνικό επίπεδο ώστε να συγκλίνουν ως προς την εξέταση προσφυγών και τις ε, διαδικασίες ενώπιν της δικαιοσύνης. Είναι η χρονιά των Ευρωπαίων πολιτών. Το 2013 όμως κάθε χρόνο πρέπει να θυμόμαστε τους πολίτες. Πολλοί λόγοι έχουν εκφωνηθεί για το θέμα αυτό, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολίτες, τουλάχιστον σε μία από αυτές τις χώρες, που θα αισθάνονται ότι πλήγονται, πλήττονται, συγγνώμη, από την έλλειψη εξέταση των προσφυγών του και την έλλειψη σχετικών διαδικασιών ενώπιον της δικαιοσύνη. Τι θα κάνετε λοιπόν εσεί γι' αυτό. Κυρία Ντανόκα. Είναι προφανές Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ε, ερώτημά μου. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Το ερώτημά μου λοιπόν προέκυψε όταν είπατε πως δεν θα μιλήσετε αγγλικά. Τι. γλώσσα την οποία μιλάτε και η δική μου γλώσσα. Είναι επίσημες γλώσσες ε, από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε πως ε, από τα 500 εκατομμύρια πολίτες δεν μιλάνε όλοι ε, τις 23 υπάρχουν ε, εκατομμύρια πολίτες που έχουν μητρική γλώσσα που δεν ανήκει στις επίσημες. Ε, αναφέρατε την, τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στα θεμελιώδη δικαιώματα και στη χάρτα αναφέρεται η απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης όταν κάποιος έχει άλλη μητρική γλώσσα. Τι θα κάνετε για αυτό το κομμάτι της χάρτας. Αν λάβετε καταγγελίες για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραδείγματος χάρη για το ότι δεν μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του, δεν μπορεί να λάβει πληροφορίες σε μια άλλη γλώσσα. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Ευχαριστώ. Mr. Ευχαριστούμε κύριο Χατζηγεωργίου. Ευχαριστώ. Ε, Γνωρίζω την κυρία Όμεν πολύ καλά ως μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών που είναι και η ίδια και ως ραπορτέρ συνακόλουθα για, για την Τουρκία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά την ευθυκρισία της, ε, την εντιμότητα της, την αντικειμενικότητα της και θέλω να τη συγχαρώ για αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλω να τη ρωτήσω μόνο το εξής. Πρόσφατα πάρθηκε μία απόφαση από το Eurogroup που ουσιαστικά λαιλάτισε τις ε, καταθέσεις ε, ανθρώπων σε μια χώρα της Ευρώπης. Εάν η ίδια ε, ήταν ή θα είναι κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας απόφασης ο Όμπουτσμαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζει ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι ή θα έκρινε ότι αυτή η απόφαση ο οπουτσμαν της ευρωπαικης ενωσης νομιζει οτι καθαρά πολιτική και δεν είναι δουλειά του Όπουτσμαν. Και η δεύτερη παρεμφερής μου ερώτηση προσωπικά κρίνω ότι οι αρμοδιότητες του Ευρωπαίου Όπουτσμαν είναι περιορισμένες. Ακόμα και αν τις συγκρίνει κανείς με τις αρμοδιότητες ενός εθνικού Όμπουτσμαν, ε, ε, στη χώρα του δηλαδή ένας Όπουτσμαν έχει περισσότερες αρμοδιότητες για την χώρα του από όσες έχει ο Ευρωπαίος ε, διαμεσολαβητής. Σκοπεύει, σκοπεύετε αν πάρετε αυτή τη θέση να προτείνετε, να σκεφτείτε, να συζητήσετε θέμα διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Martinez Martinez. Κύριε Μαρτίνες Μαρτίνες. Sí. Yo, eh, gracias, Presidenta. Yo, en primer lugar, quiero felicitar a la señora, a nuestra amiga Ría. Eh... Ευχαριστούμε την κυρία και φίλη Ρία που ήρθε και μας μίλησε στη γλώσσα της. Γιατί γλώσσα που είναι πρόεδρος Έχω και τα θέματα της πολυγλωσσίας. Αλλά εκτός από αυτό, για τη λειτουργία για την οποία θέλει να είναι υποψηφία η κυρία Ρία, η κυρία Δηλαδή, η πολυγλωσία είναι κάτι το απαραίτητο, ίσως περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στο ελληνικό μας Το να ξέρουν οι μπορούν να απευθύνονται στον ε, διαμεσολαβητή στη γλώσσα τους. Νομίζω ότι είναι σημαντικό. Είστε εδώ. Να μην το ξεχνούμε αυτό. Ότι εμείς εδώ κατευθυνθούμε και περισσότερο από Συμβούλιο και Επιτροπή πρέπει. Ακριβώς για την δημοκρατία μας ταυτότητα να θεωρούμε ότι μπορούν οι πολίτες να επικοινωνήσουν. Επικοινωνήσουν ε, ε, δεν σημαίνει μόνο απευθύνομαι, σημαίνει και γίνεται ε, αποδεκτή, ότι λαμβάνει κάποιος την πληροφορία, το θέμα το, το οποίο διαβιβάζει κάποιος. Τρεις ερωτήσεις έχω τώρα. Πρώτα πρώτα κάτι πάρα πολύ απλό. Δεν μου αρέσει καθόλου. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε ότι τη χρησιμοποιούμε για αυτή την λειτουργία κάτι το οποίο είναι ακατανόητο για κάποιον που δεν είναι Σκανδιναβός. Ombudsman, εμείς το καταλαβαίνουμε, αλλά όχι όλοι οι υπόλοιποι. Είναι ακατανόητο για τους άλλους. Γι' αυτό και λέμε διαμεσολαβητής στα ισπανικά, στα γαλλικά υπάρχει λέξη κατανοητή. Δεν ξέρω τώρα στις άλλες επίσημες γλώσσες αν υπάρχει κάποια λέξη που να ε, χρησιμοποιείται αντί για αυτήν την μυστηριώδη λέξη ombudsman που δεν λέει τίποτα για τον κόσμο. Επίσης, το πιο σημαντικό είναι η εμπιστοσύνη. Εγώ αυτό ήθελα να ζητήσω να μου εξηγήσει η προσκεκλημένη μας. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την υπόθεση εμπιστοσύνη. Αλλά επίσης πώς μπορούμε να ανοίξουμε αυτό το κοινοβουλίο, να μην γίνονται τα πράγματα εγκρυπτό και απαραβίστο, να υπάρχει εμπιστοσύνη. Γιατί μιλούμε για πάρα πολύ περιορισμένο αριθμό των συζητούντων το κάθε ζήτημα, ακόμα και όταν μιλούμε για την Επιτροπή των Αναφορών. Οπότε και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι ένας θεσμός. ένας θεσμός τον οποίο όμως αγνοεί η συντριπτική πλειοψηφία των Ευρωπαίων. Οπότε σας ερωτώ, κύριε υποψηφία, πώς νομίζετε μπορείτε να βγείτε από αυτή την κατάσταση του, του, της μυστικότητας του να μην σας ξέρει ο κόσμος. Αλλά είναι μεριά, επειδή κανεί ανοίξει πολιτικό κόμμα δεν πρέπει να αφήσετε κάποιε κυρώσει. Άλλωστε, μην ξεχνάτε ότι προέρχομαι από μια χώρα που πολιτικό κόμμα σήμαινε πα φυλακή. Μέχρι τα 37 μου ζωή σε αυτήν την κατάσταση. Όμω δεν μπορούμε κάποιον τον καταδικάζουμε επειδή ανήκει, επειδή ε, σχετίζεται με κάποιο κόμμα. Στη δημοκρατία αυτό είναι αδιανόητο. Πρόκειται για δικαίωμα, βασικό δικαίωμα του ανήκειν ει κόμμα. Αλλιώ ε, οτιδήποτε άλλο λέει κανεί, αυτό αποτελεί πλήγμα στη δημοκρατία. Πέραν αυτό τώρα θέλω να ρωτήσω την ε, φίλη μα εάν είναι υπέρ του να υπάρξει κάποιο σύστημα ούτω ώστε από πλευρά κοινοβουλίου να μπορεί ε, το, το σώμα να πάυσει από τα καθήκοντά του έναν ε, Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε και ακόμη δεν έχει διευκρινιστεί. Άρα θα πρέπει να θεσπιστεί κάποιο σύστημα, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να μπορεί να πάψει τον δημοσιογράφο. Είτε για αναποτελεσματικότητα, για έλλειψη ανεξαρτησίας κλπ. Εσείς κύριε υποψηφία, θα πάρετε τι θα παραιτιόσασταν τέλο πάντων εάν σας το ζητούσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι απλώς σας ρωτώ. Εάν το ζητήσουμε, θα ήσασταν στη θέση να παρατηθείτε. Το Κοινοβούλιο δεν έχει την αρμοδιότητα να πάψει τον διαμεσολαβητή σήμερα, αλλά έχει δυνατότητα να ζητήσει την παρατήση αυτού. Επομένω, για πετε μα, θα ήσταν θέση να παρατηρηθείτε αν το ζητούσαμε. Για έλλειψη αποτελεσματικότητα ή τέλο για εξάρτηση από συμφέροντα. Γιατί για μένα το θέμα αυτό της ανεξαρτησίας είναι πάνω απ' όλα. Εάν εγώ έχω την αρμοδιότητα να κρίνω ότι δεν είναι ανεξάρτητος ο διαμεσολαβητής, ε, τότε για μένα ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την όπω είπα, το να ανήκει κάποιο να σχετίζει με πολιτικό κόμμα. Αυτό δεν σημαίνει δεν έχει ανεξαρτησία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Τελευταίο ο κ. Μποστινάρου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μία σημαντική ερώτηση έχει να κάνει με τη δική σας υπόσχεση να φροντίσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Όλα αυτά ωραία ακούγονται, εντυπωσιάζουν, αλλά το θέμα είναι πώς θα γίνει. Η ερώτησή μου προκύπτει από το εξή. Ω σήμερα, ο Επίτροπο ή η Επίτροπο που ασχολείται με τη χάρτα, η κυρία Ρέντινγκ, αντιτίθεται στην συμπερίληψη τη Ευρωπαϊκή Χάρτας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ω ε, μέρο τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου μπορεί να μεταφερθεί μόνο στην εθνική νομοθεσία, λέει η χάρτα. Εσείς πώς προτίθεστε να το καλύψετε το θέμα αυτό της χάρτας στο μέλλον. Ε? Δεύτερη ερώτηση. Έχοντας κατά νου τη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την εμπιστευτικότητα, την έλλειψη διαφάνειας, την προστασία του παρήτου, σε σημαντικά ζητήματα, πώς θα φροντίσετε η διαφάνεια και η ταχεία εξέταση θεμάτων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα οργανωθούν στο μέλλον. Πώς? Διότι θα είναι πολύ σύντομη η θητεία σα. Δεν μπορεί να έχει πλεονάζον προσωπικό το γραφείο του Δημοσολαβητή. και του χρόνου θα έχουμε νέο, νέο διορισμό. Εκλογή και διορισμό. Πόσο τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μπορείτε να δημιουργήσετε ένα καλό θεμέλιο για μεγαλύτερη συνεργασία και διαφάνεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Επίση υπάρχει μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά των κυβερνήσεων των κρατών μελών μεταξύ του. Πώ θα διασφαλίσετε ότι τα πρότυπα που προασπιζόμαστε εδώ στι ε, Βρυξέλλε, στο Ευρωκοινοβούλιο, θα γίνουν σεβαστά και από το γραφείο του δημοσιολαβητή. Πώς θα υπάρξει συνέπεια και συμβατότητα και στη συμπεριφορά των εθνικών κυβερνήσεων. Μήπως η διαφάνεια και η καλή διοίκηση ή η κακοδιοίκηση Πώς θα διασφαλίσουμε ότι αυτά τα στοιχεία θα έχουν την ίδια, ε, ε, θα την κάνουν τις ίδιες στις Βρυξέλλες και στα κράτη-μέλη. Διότι η Επιτροπή μας θα παραμείνει ο τόπος που θα απευθύνονται οι προσφυγές των πολιτών και σαν τον πόλεμο της Ιερουσαλήμ θα μας θυμίζουν ότι οι πολίτες είναι δυσαρεστημένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι ανίκανοι να καλύψει τις προσδοκίες τους. Ευχαριστούμε κύριε Μποστινάρου. Κύριε Όμεν Ρόιτον. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με τον τελευταίο. Πώς μπορούμε να φροντίσουμε να λειτουργεί η χάρτα και στα κράτη-μέλη. αυτό θα κάνουμε και με την συνθήκη, η οποία ορίζει πως ε, ισχύει άμεσα μόνο για τα θεσμικά όργανα. Οπότε θα προσπαθήσει ο Δημοσιολαβητής, αλλά επαφείται, από το, επαφείται στο Συμβούλιο και το μετά αυτό το οποίο είπατε για μυστικότητα και διαφάνεια. Εγώ είμαι υπέρ της όσο δυνατόν περισσότερης διαφάνειας. Και αυτή είναι ακριβώς η σύγκρουση που υπάρχει. Δηλαδή, σε ποιο βαθμό μπορούμε να ακολουθήσουμε τις απαιτήσει εμπιστευτικότητας χωρίς να πληγεί διαφάνεια και θεωρώ πως μπορούμε από κοινού με το Κοινοβούλιο να ζυγίσουμε την κατάσταση για την εγγύηση της ιδιωτικότητας η οποία βεβαίω επίσης είναι πάρα πολύ σημαντική και ναι είδα 2008-2011 το τελευταίο ψήφισμα το οποίο υπήρχε αλλά Τώρα εσείς πρέπει να φροντίσετε για την νέα νομοθεσία ε, που θα συμμορφώνεται με την συνθήκη της Λισαβόνας. Επίσης, θεωρώ πως και ως κοινοβούλιο δεν πρέπει να το θεωρούμε τόσο σωστό ε, οποιαδήποτε συμβαστική θέση έχουμε εμείς στην διαδικασία της συνδιαλλαγής να υποβάλλεται στην ομάδα εργασίας του Συμβουλίου. Οπότε θα πρέπει όντως, όπως είπα, να υπάρχει η μυστικότητα και θεωρώ πως έχει καλή επαφή ε, ο διαμεσολαβητής με τα θεσμικά όργανα και μπορούμε να έχουμε και κάποια βελτίωση σε αυτό το μέτωπο. Τώρα για τον κώδικα συμπεριφοράς θα πρέπει να είναι ίδιος σε όλα τα θεσμικά όργανα. Αυτός ο οποίος υπάρχει και εφαρμόζεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ως αφετηρία τον πολίτη, ενώ ο κώδικας συμπεριφοράς, αν το συγκρίνεται δηλαδή με αυτόν του, της Κομισιόν και του Συμβουλίου, είναι γραμμένος για τον υπάλληλο και το τι πρέπει να κάνει ο υπάλληλος. Ε, πρέπει να το γυρίσουμε ανάποδα. Άρα, έτσι, να αντιστρέψουμε αυτή την κατάσταση, ε, να υπάρχει μεγαλύτερη συνεργασία και προσανατολισμός προς τον πολίτη. Πάει αυτό. Λοιπόν, επόμενο. Αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τις καταθέσεις. Πρέπει να το σκεφτώ, αλλά θεωρώ πως έτσι, πρώτης όψεως, δεν μπορεί να κάνει τίποτα ο πολίτης. Ο πολίτης πρέπει να απευθυνθεί στον νομοθέτη στη χώρα του. Και εκεί πέρα ο διαμεσολαβητής, αλλά ο δικός σας διαμεσολαβητής ε, ε, έχει νομίζω κάποιο ρόλο, αλλά αντιλαμβάνομαι το, το πρόβλημα. Τώρα, πώς θα μπορέσουμε να συνεισφέρουμε έτσι ώστε να αποκτήσουν όλες οι χώρες δημοσιολογητή. Ε, δεν μπορούμε να το απαιτήσουμε, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε και με όλα τα κράτη-μέλη, με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα κράτη-μέλη για να υπάρχει και εκεί πέρα ένα τέτοιο θεσμικό όργανο. Συζητήματα στα οποία είχα εργαστεί σε θέματα διεύρυνσης ε, ζητούσαμε αν είναι δυνατόν να υπάρξει και ε, διαμεσολογητής. Κατόπιν κύριε Μαρτίνη σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Η πολυγλωσία είναι σημαντική πράγματι. Αυτό δεν σημαίνει όχι μόνο και για την υποβολή ενός αιτήματος αλλά και για την απάντηση. Εδώ πέρα συμφωνώ 100% αλλά και εδώ πέρα απευθύνομαι και στην κυρία Σαντονόκα. Αυτό σημαίνει πως τη στιγμή κατά την οποία τα ρώσικα δεν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πολίτης ε, δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα ρώσικα σε ένα επίσημο αίτημα προς τον διαμεσολαβητή. Ε, αυτά προβλέπει η συνθήκη. Έτσι, ε, και πρέπει να συμμορφωθεί ο διαμεσολαβητής. Οπότε για τα γλωσσικά μην ανησυχείτε. Ε, με μένα είναι σε καλά χέρια. Ο εσείς λέτε Defensor de Pueblo, οι Γερμανοί λένε Bürger Beauftragte, στην υπηρεσία του πολίτη δηλαδή. Και νομίζω πραγματικά το αντικατοπτρίζει καλύτερα την ουσία αυτής της υπηρεσίας. Και αυτό που λέτε εσείς, ε, συνήγορος του πολίτη, υπερασπιστής του πολίτη, κάποιος ο οποίος έχει εντολή να υπερασπίζεται τους πολίτες από ε, τη διοίκηση. Αλλά η λέξη Ombudsman είναι μία λέξη, δεν ξέρω, νομίζω σκανδιναβική. Απευθύνομαι στην κυρία Άουκεν, κάπου εκεί από τη Σουηδία, Φιλανδία, Δανία. Α, δεν έχω κάποιο πρόβλημα με τη, λέξη τώρα, δεν είναι θέμα. Πώς θα πρέπει τώρα να λειτουργεί η Μεσολαβητής αυτό το πρέπει να κάνει ο ή μεσολαβητή είναι να αυξήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Να δούμε πώς ως εντολοδόχος των πολιτών ε, μπορεί να αποκαταστήσει την ε, εμπιστοσύνη και να είναι προσανατολισμένος προς τους πολίτες και όχι προς τα θεσμικά όργανα. Και προς αυτήν την κατεύθυνση θέλω να εργαστώ και θεωρώ πως μία από τις ικανότητες που έχω είναι η πειθό το να ε, ρίχνω γέφυρες, δηλαδή προς άλλους και έτσι να α, ε, μπορέσω να μεταπίσω τα θεσμικά όργανα. Μετά υπήρχε ένα πολύ ε, συγκεκριμένο ερώτημα, αν μπορεί να απολυθεί ο διαμεσολαβητής. Ναι, ναι, βεβαίω. Ε, ελπίζω να μην γίνει, αλλά αν πραγματικά το Κοινοβούλιο θεωρεί πως ε, υπάρχει παραβίαση του τρόπου λειτουργίας κτλ. Πρέπει να το κάνει και αναφέρεται στην συνθήκη. 10% των βουλευτών μπορεί να κάνει μια πρόταση για την απόλυση του δημοσιολογητή. Έτσι. Κατόπιν. Κύριε Χατζηγεωργίου. Είπατε πράγματι πως ε, έχω τις σχετικές εμπειρίες από την πολιτική και τα λοιπά. Σας ευχαριστώ. Μετά ο κύριος Μπουλόν. Δεν έχει κάθε κράτο μέλος ε, διαμεσολαβηθεί πράγματι. Πώς μπορώ λοιπόν να ρίξω το βάρος μου για να αποκτήσει το κάθε κράτος μέλος διαμεσολαβηθεί. Πρέπει να γίνει η δουλειά με τα θεσμικά όργανα που υπάρχουν σε κάθε κάτω μας. Αλλά η χάρτα πρέπει να εξαπλωθεί νομίζω, αυτό είναι το σημαντικότερο. Αλλά δεν έχω καμία ε, δυνατότητα τυπική ε, να υποχρεώσω κάποιον όπως είπα προς αυτή η κατεύθυνση. Αυτά νομίζω. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ολοκληρώσαμε τις ακροάσεις για σήμερα το πρωί. Οπότε ευχαριστήσω προς όλους. Ιδίως προς την κυρία Ρόιτεν και της εύχομαι καλή τύχη. Σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε το απόγευμα.